Colleagues, once more, please be seated. Συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ, λέει η πρόεδρος. I'm sorry for this long... Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση, λέει η πρόεδρος της απογευματινής συνεδρίασης. Τώρα είμαστε πλέον καθόλου έτοιμοι. Έχουμε εδώ μια πολύ σημαντική ενημέρωση από τον κύριο Πασκού σχετικά με το πρόγραμμα ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανίας, την πρόταση και την εκκίνηση του τριμερούς διαλόγου. Ο ο κύριος Πάσκου έχουμε ένα τέταρτο περίπου για την ενημέρωση αυτή. Παρακαλώ τον εισηγητή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι πράγματι ο πιο σημαντικός, όπως είπατε πρόεδρε, διαθέσιμος. Να μην πούμε ότι είμαι και ο πιο σημαντικός δηλαδή, είμαι απλά ο διαθέσιμος. Είχαμε λοιπόν κάποιες επαφές ήδη από το Στρασβούργο εν ώψη του τριμερούς διαλόγου, μάλλον μία συνάντηση τριμερούς διαλόγου, μία τεχνική επίσης συνάντηση στα πλαίσια αυτά, και πάνω κάτω σε σχέση με τα τέσσερα σημεία υποσυζήτηση δεν υπήρξε ιδιαίτερη κίνηση. Αυτά τα τέσσερα σημεία έχουν σχέση με τον προϋπολογισμό, μη επιλέξιμες δράσεις, επιλέξιμες οντότητες και πρόγραμμα εργασίας. Βρήκαμε κάποια συμβιβαστική ορολογία επί ενός και μόνο σημείου τα συστήματα δηλαδή που διανόμου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται. Έχουμε συμφωνίες, έχουμε ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, θέλαμε μια σαφή και ρητή μία. Στην ουσία λοιπόν αυτά τα έχουν αποδεχθεί Συμβουλίο και Κομισιόν. Αυτή τη συνταγή επί της αρχής την έχουν αποδεχθεί. Τώρα όταν επί παραδείγματι μιλούμε για επιλέξιμες οντότητες, το Συμβούλιο έχει κάποιες ιδέες ότι εφόσον υπάρχει εγγύηση για το κράτος, τότε θα πρέπει να είναι αποδεκτό. Εμείς στο Κοινοβούλιο θέλουμε περισσότερες εγγύησεις. Για να σας δώσω μία εικόνα για τα σημεία τα πιο δύσκολα. Στην τεχνική τώρα συνάντηση εχθές μου ελέγχθη διότι δεν επιτρεπόταν η συμμετοχή μου μετεφέρθη λοιπόν μια δυσάρεστη ανταλλαγή υπάρχουν έχει βιντεοσκοπηθεί πώς λοιπόν μεταχειρίστηκαν τους δικούς μου ανθρώπους, τους δικούς μου βοηθούς, η υπεύθυνη ασφαλεία. Έχω γράψει σχετικά με το θέμα στον κύριο Μπούζε και στον κύριο Ταγιάννη, καταγγέλλοντα το περιστατικό και διαμαρτυρώμενο σχετικά, αλλά πέραν αυτού, όπως με ενημέρωσε η γραμματεία, η συζήτηση δεν οδήγησε στην εξέβρεση κοινού εδάφους. Πάντως θα έχουμε επόμενο τριμερή διάλογο 10 Απριλίου και δύο-τρεις τουλάχιστον ακόμα τεχνικές συναντήσεις. Υπάρχει λοιπόν μια δυνατότης, μια πιθανότης για άλλον έναν τριμερή στο τέλος Μαΐου εφόσον δεν βρεθεί κοινό τόπος νωρίτερα. Όλα αυτά δεν είναι ξαφνικά ή ανευπροηγουμένου, είναι λίγο ως πολύ κανονικά ως προς το πώς εξελίσσονται αυτές οι συζητήσεις των τριμερών διαλόγων προκειμένου να βρεθεί ένας κοινό τόπος για την ε, κίνηση της πρωτοβουλίας του χρόνου διότι το χρονοδιάγραμμα είναι εξαιρετικά επιβαρημένο εμείς το τηρήσαμε ως κοινοβουλίο Αυτά είχα να σας πω πρόεδρε, ευχαριστώ. Μάλιστα, ο κύριος Άρνολς, παρακαλώ, ευχαριστώ πρόεδρε. Είχαμε σε άλλες συναντήσεις θέση το θέμα των κοινών σημείων, τα οποία θα ήθελα να υπογραμμίσω για το πού βρισκόμαστε δηλαδή στην χρηματοδότηση και εν ώψη των συζητήσεων του ΠΔΠ Επίσης τα κονδύλια, οι τίτλοι των κονδυλίων χρησιμοποίησης βιομηχανικής ανάπτυξης θα πρέπει να βρεθούν από υφιστάμενα προγράμματα και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμπληρώσουν Και ως προς το χρονοδιάγραμμα πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να φοβηθούμε να απαιτήσουμε περισσότερο έλεγχο κοινοβουλευτικό, διότι πρέπει να είμαστε μια πλήρης επιτροπή στο μέλλον, να έχουμε κοινοβουλευτικό λέγειν και έλεγχο. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε στενά συνδεδεμένοι με την όλη αυτή διαδικασία, για την έρευνα, για τις αποφάσεις για τις εξαγωγές, για τα αμυντικά συστήματα, ιδιαίτερα σε σχέση με την ενωσιακή χρηματοδότηση, που δεν θα είναι αναγκαστικά σημεία προτεραιότητα σε αυτό το τριμερή διάλογο, αλλά πρέπει να λάβουμε μια ευρύτερη εικόνα, μια ευρύτερη προοπτική για να προχωρήσουμε επί αυτών. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κ. Δροϊεύσκη. Chcę bardzo serdecznie podziękować panu Pasku. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Πάσκου γιατί κατανοώ το μέγεθος των δυσκολιών που δεν αφορούν μόνο τις ρυθμίσει του τριμερούς διαλόγου αλλά και τις συζητήσει με τις άλλες επιτροπές. Να μην ξεκινήσουμε τώρα μια συζήτηση για την έκθεση γιατί ήδη έχουμε δώσει την εγκρισή μας. Όμως έχω κάποια επιμέρους ζητήματα να σχολιάσω. Να ρωτήσω καταρχάς τι γίνεται και σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε σε σχέση με τον εντοπισμό αυτών που συλλογικά ετούνται αυτούς τους δημοσιονομικούς πόρους. Μετά, για τα ποσά. Ποια είναι η διαφορά η απόκληση μεταξύ αυτών που συζητάμε εμείς και αυτών που έχουμε σήμερα μπροστά μας διαθέσιμα. Και κατά πόσο όλα αυτά σχετίζονται με τις προηγούμενες συζητήσεις μας που είχαμε νωρίτερα δηλαδή για την κυβερνοασφάλεια. Στην έκθεσή σας εσείς παρουσιάζετε νομίζω σωστά τις υβριδικές απειλές και την ανάγκη να επεκταθούμε στα θέματα ασφαλείας και στην κυβερνοασφάλεια. Υπάρχουν εδώ στοιχεία τα οποία μπλέκονται και για το δεν υπάρχει συμφωνία ή υπάρχει πλήρης ε, ομόνια. Ευχαριστώ λέει πρόεδρο και εγώ θα προσθέσω και δύο ερωτήσεις σε αυτέ που ανέφερε ο κύριος Στριεύσκη, δύο δικέ μου δηλαδή ερωτήσει, λέει πρόεδρο, σε σχέση με τον αριθμό των οντοτήτων. Συμφωνώ απόλυτα με την άποψη ότι πρέπει να είναι πάνω από δύο, όμως θα ήθελα να πω επίσης ότι και η θέση ή η σημασία των μεσαίας κεφαλαιοποίησης ή οικονομικής ευρωστίας επιχειρήσεων και αυτή σημαντική, ιδιαίτερα από υπερατλαντική σκοπιά για τον ΝΑΤΟ και για άλλους τομείς. Πρέπει να υπάρχουν λοιπόν κάποιες διατάξεις που διασφαλίζουν την συμμετοχή και τρίτων χωρών τουλάχιστον για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Με την εξαίρεση βέβαια χωρών που έχουν θέση επιθετική, να το πω κάπως λέει ο Πρόεδρος. Α, δεν ξέρω τι γίνεται. Κύριε Πασκού, έχετε το λόγο. Για πείτε μας. Ναι. Περισσότερα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την άμυνα σημαίνει περισσότερη δυνατότητα αποπτίας για το κοινοβουλίο μας, δηλαδή αυξημένος ρόλος του κοινοβουλίου. Θα δούμε μετά βέβαια κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Θα δούμε στο μέλλον. Τώρα, για τις εξαγωγές, η πρωτοβουλία αυτή δεν αφορά τις εξαγωγές. Δηλαδή, δεν αποτελεί ένα παραθυράκι για να επαναθήξουμε το θέμα το οποίο έχει ρυθμίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή εξαγωγές όπλων. Οπότε το θέμα των εξαγωγών επαφείται καθαρά στις χώρες μέλη. Το Συμβούλιο ζήτησε και φοβάμαι ξέρετε ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε περισσότερη νομοθεσία για τις εξαγωγές όπλων μέσω παραθύρων όπως αυτή εδώ η νομοθεσία. Για το και η ΣΕΝΤΕ και η ΤΡΕ και στον τριμερή διάλογο υπόθηκε ξεκάθαρα. Δηλαδή, εγώ δεν έντοψα κάποια διαφωνία εκ μέρους Συμβουλίου Κομισιόν για αυτό το θέμα και φαντάζομαι στο τέλος θα περάσει. Τώρα, για τον προπολογισμό, εντάξει, νέα κονδύλια, αλλά τι γίνεται με τα κονδύλια τα οποία δεν έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε άλλα προγράμματα. Δόθηκαν στο, παλαιό, στο παρελθόν, συγγνώμη, είναι παλιά κονδύλια, οπότε δεν εμπίπτουν εδώ ή είναι ελεύθερα κονδύλια, οπότε θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν. Δεν ξέρω πώς θα το ερμηνεύσουμε αυτό, αλλά βεβαίως θα το συζητήσουμε όταν θα μιλήσουμε για την έκθεση των, που αφορά τη σχέση μεταξύ που αφορά την Ένωση και το ΝΑΤΟ. Είναι στα πλαίσια του θεματολογίου μας, θα υπάρξει νομίζω κάποια καλή συνεργασία. Τώρα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μεσαίες κεφαλαιοποίησεις επιχειρήσεις. Είχαμε κάτι, αλλά αφαιρέθηκε και υπάρχουν δύο όροι, από ό,τι ξέρω που χρησιμοποιούνται μαζί, που περιγράφουν δηλαδή δύο κατηγορίες. Αυτή η λύση δηλαδή καλύπτει δύο περιπτώσεις. Μικρομεσαίες, αλλά και πιο κεφαλαιοποιημένες που είναι επιλέξιμες. Για τις τρίτες χώρες τώρα υπάρχουν κάποια πράγματα που αναπόφευκτα τις εμπλέκουν και θα συνεχιστεί αυτό. Όμως καταλαβαίνω την άποψη του κυρίου Νταντζάν που διατύπωσε εδώ και καιρό και λέει ότι και άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν ε, μάλλον ρωτάει, έχουν υποφελήθει κονδυλίων στις ΗΠΑ ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Δεν έχω απάντηση γι' αυτό. Μάλλον έχω, αλλά θέλω να την πω δημόσια. Ιδιαίτερα τώρα, μια και βρισκόμαστε στην αρχή και θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε το κοινό για αυτή την αλλαγή στο υπόδειγμα, με βέβαιος ότι θα βρούμε μια λύση. Κάποιοι προτείνουν τα προγράμματα της ΠΕΣΚΟ να μην αποκλείουν χώρες όπως η Βρετανία μετά το Brexit ή η Νορβηγία, ξέρω εγώ, να συμμετάσχουν αν όντω θέλουν να έχουν ενεργό συμμετοχή. Το λέω αυτό για παράδειγμα. Δεν ξέρω αν θα συμβεί ή όχι, αλλά τέλος πάντων αναφέρθηκε και αυτό ως ιδέα. Θα θέλαμε λοιπόν να το αφήσουμε ανοιχτό όσο γίνεται για τις τρίτες χώρες. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τον άλλο παράγοντα, ότι δηλαδή αυτή η πρωτοβουλία είναι νέα και είναι αντικείμενο συζήτηση το τι σημαίνει αυτόνομη στρατηγική. Υπάρχουν ορισμοί γι' αυτό και θεωρώ ότι στα πλαίσια της έκθεσης για να μην υπάρχουν επίμαχα ζητήματα μιλάμε μόνο για την διατήρηση της αυτονομίας λήψης αποφάσεων. Στην έκθεση αναφέρω αυτούς τους δύο οργανισμούς, στον οποίο η δυνατότητα λήψης αποφάσεων θα πρέπει να είναι σεβαστή και μετά θα δούμε για τους υπόλοιπους οργανισμούς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. για όλες αυτές τις ε, παρατηρήσεις, αλλά θα ήθελα να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα, γιατί πραγματικά ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε σας ζητώ συγγνώμη κύριε Γκάλερ, μπορείτε να παρέμβετε τώρα και μετά συνεχίσουμε. Ναι. Απαντώντας τον Άννα και υποστηρίζοντας τα όσα είπε ο Σάνθος Απάσχο, αυτό το EDP είναι ακριβώ για την περίοδο 2019-2020 έω δηλαδή να φτάσουμε στο επόμενο το δημοσιονομικό πλαίσιο. Άρα λοιπόν η συζήτηση ω προ τι δαπάνε και στο ύψο του αφορά στο επόμενο ε, πλαίσιο. Θα πρέπει δηλαδή να, σε αυτό το πλαίσιο να εντοπίσουμε ποιε είναι οι προτεραιότητές μας και τι χρειαζόμαστε για αυτές τις προτεραιότητες. Δεν θέλω δηλαδή να πάρω κονδύλια από το Horizon για παράδειγμα για να τα κατευθύνω αλλού και δεν θέλω για παράδειγμα να υπάρξει μια διαμάχη ή ένα ανταγωνισμό αν θέλετε μεταξύ ερευνητών και αγροτών ε, ε, για παράδειγμα και το μέτρη μήνας αφετέρου. Θέλουμε λοιπόν ε, να είμαστε θαραλέοι και να δούμε ποιε είναι οι πολιτικέ τι οποίε θέλουμε να προωθήσουμε και να προσαρμόσουμε ε, τη χρηματοδότηση ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες. Πάντως, σε ό,τι αφορά τον τομέα της άμυνας, πραγματικά υπάρχει εδώ μια διαφυσβήτητη ανάγκη για περισσότερη χρηματοδότηση, καθώς χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία σε αυτό το τομέα. Και μέχρι στιγμής τουλάχιστον είμαι σίγουρος ότι θα το επιτύχουμε. Δηλαδή, ε, στο, στην τελευταία φάση των ε, διαπραγματεύσεων ε, για, τον, για τη σχηματισμό κυβέρνηση συνασπισμού στη Γερμανία υπήρξε μια συζήτηση σε ό,τι αφορά τους ερευνητές και όσους ήταν από το τομέα της άμυνας υπήρξε το επιχείρημα που υπόθηκε ότι για το ένα ευρώ που επενδύεται στην έρευνα επιτυχαίνουμε κάτι αντίστοιχο στο τομέα της άμυνας. Νομίζω πως είναι ίδια η συζήτηση εδώ. Δηλαδή μέσω της αναπτυξιακής ε, συνεργασίας, μέσω της ανθρωπιστικής ε, ε, υποστήριξης πάμε στον τομέα της αμήνας μέχρι για παράδειγμα και στην αγορά αεροσκαφών πολεμικών. Οπότε Εντάξει, εσείς διαπραγματευτήκατε με την Προεδρία του Συμβουλίου, αλλά είχατε μία εντύπωση ως προς το ποια είναι η τοποθέτηση των διαφορετικών κρατών μελών με αυτό το ζήτημα. Κύριο Σπάσου. Ναι, όχι, δεν έγινε λεπτομερή συζήτηση. Απλώς η Προεδρία παρουσίασε κάποιες βασικές τοποθετήσεις από την πλευρά του Συμβουλίου. Δεν ξέρω αν υπάρχει ομοφωνία δηλαδή στο Συμβούλιο. Κύριο Εάν υπάρχει μια πολύ σημαντική επιχείρηση στην, ε, στην ε, Γερμανία, η οποία έχει ε, την νομική έδρα και είναι εταιρεία περιορισμένη σε αυτήν στη Γερμανία, η οποία βέβαια είναι Αμερικανικών συμφερόντων και η οποία αρμόδια για τον έλεγχο σε ακτίνες δηλαδή των αποσκευών. Και σε σχέση με μια άλλη επιχείρηση, για παράδειγμα, υπήρξε δυνατότητα στο πλαίσιο του Brexit ότι θα μπορούσε να γίνει μια μεταγκατάσταση ε, στι ΗΠΑ, με αντίστοιχη επιχείρηση. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι κάποιες ε, από αυτές τις επιχειρήσεις, ε, εφόσον ε, το δικαιούνται, θα αναλάβουν τα στηριότητα αυξημένα εδώ στην υπηρετική Ευρώπη. Και σε ό,τι αφορά τώρα τα project τα οποία αναφέρθηκαν, δεν θέλουμε τρία συν τρία όπως αναφέρθηκε, αλλά παραπάνω. Πρόεδρο, ο κ. Δεζόν θέλει να παρέμβει. Καλώ, θα του δώσουμε το λόγο, αλλά παρακαλώ πολύ σύντομα γιατί έχουμε καθυστερήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε απλώς σε σχέση με τα όσα έλεγε ο κύριος ε, Πάσκου ε, σχετικά με την τοποθέτηση που είναι αρκετά ε, αυστηρή αν θέλετε από αυτού το γεγονό ότι τρίτες χώρες και μάλιστα πολύ περισσότερο σύμμαχες χώρες να μπορούν να συμμετάσχουν στα πράγματα συνεργασίας είναι απολύτως θεμητό. Το ζήτημα είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια Δηλαδή η συμμετοχή δεν πρέπει να σημαίνει κατά ανάγκη και χρηματοδότηση. Και έχω ακούσει από σημαντικές προσωπικότητες Ευρωπαίους ότι ευρωπαϊκά προγράμματα θα μπορούσαν να σηματοδοτούν, να διαδραματίζουν, να σημαίνουν ένα κίνδυνο στο θέμα των ατλαντικών σχέσεων. Αλλά ε, δεν ισχύει κάτι τέτοιο γιατί δεν μπορεί να με πείσει κανείς ότι η αμερικανική βιο... Ε, αμυντική βιομηχανία και στις διεθνείς της ε, θα μπορούσε να απειλείται από ένα πρόγραμμα τόσο μικρό όσο αυτό που συζητούμε. Δεν είναι ένα δισεκατομμύριο που θα απειλήσουν την ε, αμερικανική αμυντική βιομηχανία. Δηλαδή ας είμαστε ε, σοβαρή. Επομένως νομίζω ότι πρέπει να διακρίνουμε τα πράγματα συνεργασίας ε, με τρίτες χώρες αλλά να έχουμε κατά νου και τους όγκους τους σχετικούς. Μάλιστα λέει η Πρόεδρος, νομίζω ότι εδώ θα έπρεπε να ολοκληρώσουμε με το σημείο αυτό της μισής διατάξεως το οποίο κράτησε λίγο περισσότερο από ό,τι είχαμε προβλέψει για να πάμε τώρα την πρώτη εξέταση του σχεδίου εκθέσεως για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Η είναι ο κ. Πάσχου. Η 28 η Μαρτίου είναι η προθεσμία της υποβολής των τροπολογιών. Κύριε Πάσκου, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, η έκθεση είναι έτοιμη και νομίζω ότι γνωρίζετε κι εσείς ότι υπάρχουν τρεις βασικοί αξονές, τρία σκεπτικά πριν των οποίων ε, δομείται η έκθεση αυτή. Ότι πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ είναι απολύτως φυσιολογικοί σύμμαχοι. Έχουν ίδια στόχευση, και επομένω πρέπει να συνεργάζονται. Δεύτερον, η συνεργασία που είχαμε τελευταία χρόνια είναι ακόμα στο ξεκίνημά της, θα λέει κανείς, λέει ο μιλητής. και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε άλλη μια διακήρυξη τον Ιούλιο Ευρωπαϊκής Ένωση ΝΑΤΟ σχετικά με τη συνέχιση της συνεργασίας αυτής που θα περιλαμβάνει και περισσότερες ε, αν θέλετε πτυχές και τρίτον έχουμε αρχίσει να ασχολούμεθα σοβαρά με σημαντικά ζητήματα όπως είναι οι μεταφορές. Το δίκτυο, το μεταφορικό είναι ε, ισοδύναμο με την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί μέσω αυτής δομηθική ακόμα βεβαίως προσανατολίζεται από Ανατολάς προς Δυσμάς δεν έχουμε στον βορειο-νότιο άξονα κάτι ιδιαίτερα προς τις ανατολικές περιοχές και κάτι που θα πρέπει να κάνουμε αλλά μας ενθαρρύνει το έργο που έχει ήδη ξεκινήσει η EDA έχει ήδη αφιερωμένη σε αυτό ομάδα και η οποία είναι πολύ επιτυχής μέχρι στιγμής στην ενέργειά της, στην προσπάθειά της, αλλά θα κλείσω λέγοντας ότι η πραγματική δοκιμασία των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ είναι τι θα κάνουν σε περίπτωση κρίσεως στην Ευρώπη. Όχι αλλού, στην Ευρώπη. Δεν μιλάω για τον Βόρειο Ατλαντικό ή κάπου αλλού, μιλάω για το ευρωπαϊκό έδαφος. Εν πάση η έκθεση γύρω από αυτά τα σημεία του μύτη. Και άπτητε και επικοινών απειλών και προκλήσεων και περιοχών στις οποίες κατέχουμε μία αριστεία θα έλεγα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ όπως και επί των όσων κάνουμε από κοινού για τις υβριδικές απειλές τις απειλές του κυβερνοχώρου παραδείγματος χάρη γνωρίζω ότι εκεί ε, μεταχειριζόμαστε Κάποιε φορέ ελαφρώ διαφορετικά κριτήρια, καλό θα ήταν να χρησιμοποιούμε τα ίδια κριτήρια. Από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ είναι σημαντική ιδίως για τη σχέση τη δική τους με τον ΝΑΤΟ περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η φυστάμενη κυβέρνηση θα ήθελε κάποιες εγγυήσει ότι τα όσα κάνουμε εδώ δεν είναι επιζήμια ή δεν θα μπορούσαν να είναι επιζήμια προς τα αμερικανικά συμφέροντα ή τις διατλαντικές σχέσεις. Μερικές φορές αντιλαμβανόμαστε μια τοποθέτηση σε άξονα Νορβηγίας και Ηνωμένου Βασιλείου σε παρένθεση Brexit. Μερικές φορές έχουμε την αίσθηση ότι εμπιστεύονται περισσότερο τους Νορβηγούς και τους Βρετανούς και πάλι σε παρένθεση Brexit. Αλλά δεν μπορεί το ΠΕΣΚΟ να είναι μια υποενότητα, δηλαδή αν κανείς λαμβάνει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν, το, λαμβάνει χρηματοδότηση από τον ΝΑΤΟ, τελικώς θα χρησιμοποιήσει το ίδιο πρόγραμμα που θα πρέπει να είναι υποφελές για όλους. Τώρα στα πλαίσια του Neighbors and Partners, γείτονες και σύμμαχοι, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια αυξημένη ανθεκτικότητα για τους εταίρους μας, λέει ο Μιλτής. Τώρα να πω ότι 19 Μερτίου ο Γενικός Γραμματέας ε, ε, εξέδωσε την ετήσια έκθεσή του. Την έχω διατρέξει, έχει τμήματα που αναφέρονται στη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έλεγα για τις υβριδικές απειλές, τις ε, απειλές του κυβερνοχώρου, τα ζητήματα μεταφορών, Όλα αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά για το μέλλον των σχέσεων μεταξύ των δύο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα μιλήσω ως Κιώδης, αλλά εξ ονόματός μου. Συζητήσαμε πάντως με τον εισηγητή για θέση της ομάδας. Ευχαριστώ τον κύριο Πάσκου για αυτό το αξιόλογο εγγραφό που προσδιορίζει τους κυρίους τομείς συνεργασίας. Δεν θα αναφερθώ στα θετικά, αλλά στα προβληματικά σημεία. Καταρχάς, θα πρέπει να αναφερθούμε στο ότι δεν έχουν να κάνουν με τους ίδιους οργανισμούς και δεν έχουν τη διαφύση αυτοί οι οργανισμοί. Εγώ βλέπω στο κείμενο αυτό να επιμένουμε ίσως υπερβολικά για την ταυτότητα, στρατηγική ταυτότητα, ταυτότητα απόψεων, την κοινή αυτών των οργανισμών. Είναι αλήθεια υπάρχει, αλλά δεν μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Μιλάμε για μια στρατιωτική συμμαχία, πολύ συγκεκριμένη, έστω και αν περιλαμβάνει πολλά μέλη της Ένωσης, αφενός και αφετέρου την ίδια την Ένωση, την Ευρωπαϊκή, που είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, πολιτικής φύσης, που παρουσιάζει ένα εγχείρημα πολύ πιο ευρύ από ό,τι μια στρατιωτική συμμαχία. Υπάρχουν λοιπόν σημεία όπου επανειλημμένως αναφέρεται ότι υπάρχει ταύτιση στόχων και απόψεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Εντάξει, είναι αλήθεια αυτό σε κάποιου τομεί για την άμυνα και την αντιμετώπιση των απειλών, αλλά αυτό αφορά κυρίως το ΝΑΤΟ. Και ιδιαίτερα, αν δούμε τι γίνεται στο κυβερνοχώρο και στις απειλές, εγώ θα έλεγα ότι δεν θα έπρεπε τόσο εύκολα να έχουμε αυτό το κομμάτι, το σκέλος ε, του κυβερνοχώρου και της ικανότητά του να το αφήνουμε στο ΝΑΤΟ. Ε, εντάξει, το ΝΑΤΟ μπορεί να είναι πιο μπροστά, μπορεί να έχει περισσότερη ικανότητα, ας πούμε, στρατιωτική κυβερνοπροστασίας. Όμως οι κυβερνοαπειλές είναι πολύ πιο ευρειε από αυτό. Όλη η δουλειά που έχει γίνει για την κυβερνοασφάλεια, την ε, ε, το πόσο ευάλωτοι είμαστε στο κυβερνό χώρο. Εντάξει, όλα αυτά στη χώρα μας πούμε, βεβαίως έχουν να κάνουμε το ΝΑΤΟ, όμω δεν απαραίτητα αυτή η μόνη οδό. Εντάξει, να υπάρχει συνεργασία, ναι, να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων, ναι, αλλά να προσέχουμε έτσι, μην έχουμε μια υπερβολική σύγκληση σε τομεί όπου θα πρέπει να διατηρηθεί η αυτονομία και η ιδιαιτερότητα του κάθε οργανισμού. Επίσης, για τα ευρυδικά και τα θέματα του κυβερνοχώρου. Το ευρυδικά εμένα δεν μου αρέσει και τόσο. Και μάλιστα ένας προλαλής εδώ είχε πει ότι υβριδικό αποτελεί ένα ορισμό και ένα όρο νέο που χαρακτηρίζει πραγματικότητες και αταστάσεις οι οποίες είναι παραδοσιακές, κλασικές. Εντάξει, ωραία αυτή η όρη, αλλά δεν χρειάζεται να επιμένουν υπερβολικά για αυτέ τις νέε καταστάσεις, για να είναι και τόσο νέε. Πέρα από τη μασμισολογία λοιπόν του υβριδικού, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το θέμα, το στρατιωτικό άμυνα, το οποίο δεν προποθέτει άμυστα αυτή με το ΝΑΤΟ. Γιατί υπάρχουν, θεωρώ, τομεί όπου υπάρχουν ιδιαιτερότητε πολύ πιο ευρείε, πολύ πέραν του ΝΑΤΟ δηλαδή. Δυστυχώ, επειδή το ΝΑΤΟ έχει μια ικανότητα μεγαλύτερη και αυτομάτως κάνουμε κάποια πράγματα μαζί προς τα εκεί προστρέχουμε αλλά νομίζω θα πρέπει να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση εδώ ιδιαίτερα στα θέματα στρατιωτικά νομίζω θα πρέπει επίση να προσέχουμε και να είμαστε προσεκτικοί για τι φιλοδοξίε όσον αφορά τη συνεργασία μα. έχουμε ένα κείμενο το οποίο σε σχέση με την Βασοβία είναι πολύ φιλόδοξο καταγράφει 40 τομεί όπου έχουμε τα κτλ. Όμως, αν δούμε τον απολογισμό σήμερα, υπάρχουν ακόμα πολλά πρέπει να γίνουν για αυτά τα 42 σημεία, έτσι. Να μην το παρακάνουμε, λοιπόν. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε και άλλα θέματα. Μετά τη Βαρσοβία, θέλουμε να προσθέτουμε και άλλα συνεχώ και αυτό δεν νομίζω να συνετώ. Και κάτι τεχνικό. Εγώ έχω αμφιβολίες σε σχέση με την επαναδιαπραγμάτευση του Βερολίνο Plus το Βερολίνο Plus είναι κάτι το πολύ συγκεκριμένο, το πολύ ιδιαίτερο, το οποίο δημιουργήθηκε σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο πριν από 15 χρόνια. Και δεν είμαι βεβαίω ότι σήμερα ε, είναι θέμα προτεραιότητας για αναθεώρηση του Βερολίνου ΣΥΝ. Και ιδιαίτερα αν έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει πάντα αυτή η φιλοδοξία του ΝΑΤΟ να αναπτύξει το αστικό, το πολιτικό μάλλον κομμάτι. Οπότε Για μένα αυτή, αυτό δεν είναι θέμα προτεραιότητας ή το πολιτικό σκέλος και αναπτυξή του από τον ΝΑΤΟ. Αυτά είχα να πω. Πάντως υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία στην έκθεση και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να τονίζουμε συνέχεια ότι δεν μιλάμε για οργανισμούς που έχουν ταυτόσημη φύση και ότι αυτόματα δεν υπάρχουν θέματα που από ένα στον άλλο. Ευχαριστώ ο κύριος Βανόλτερ, ως και όλες τις από την πλευρά του ECR. Θέλετε το λόγο? Όχι, ευχαριστώ. Κυρία Πάουτμαντς. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Πάσκου για τη δουλειά του εδώ. Όπω ε, και οι συνάδελφοι από το ΕΛΚΑ, ε, θεωρούμε πως αυτό το έγγραφο σε ό,τι αφορά τα βασικά του σημεία είναι σωστό καθώς ε, πράγματι το ΝΑΤΟ εδώ και πολλά χρόνια έχει φροντίσει για την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα όμως οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ξεκινούμε τις εργασίες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς μια Ευρωπαϊκή Ένωση Άμυνας. Και αυτό σημαίνει ότι οι εν λόγω θα πρέπει να επιταθούν και να επιταχυνθούν. Σε ό,τι αφορά αυτή την έκθεση για τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, θα πρέπει να τονίζουμε ότι η συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εξίσου σημαντική με τη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ βρισκόμαστε στην ίδια κοινότητα αξιών και χρειάστηκε πολλές φορές να ζητήσουμε για τα τελευταία χρόνια από το ΝΑΤΟ υποστήριξη. Και θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονε απέναντι στο ΝΑΤΟ για αυτήν τη βοήθεια που μα έδωσε. Υπήρξε ένα μεγάλο σύμμαχό μα και θα πρέπει σε αυτό το πλαίσιο να τονίσουμε ορισμένα στοιχεία τα οποία ενδεχομένω να επαναλαμβάνω και τα οποία ενδεχομένω ήδη να περιλαμβάνονται στην έκθεση. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να τα τονίσω. Καταρχήν, τα χημικά, βιολογικά και ε, πυρηνικά όπλα είναι ένας ε, τομέας στον οποίο θα πρέπει να συνεχίσουμε την ε, δική μας συνεργασία. Γνωρίζουμε δηλαδή ότι υφίστανται εδώ απειλές και δεν α, τις παραγνωρίζουμε. Γνωρίζετε ε, κυρία Πρόεδρε, πω υπήρξε μια έκθεση πρωτοβουλία από τη δική μου πλευρά ω προ το πώ μπορούμε να συνεργαστούμε και με τον ιδιωτικό τομέα σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Και εδώ ίσως θα πρέπει να το τονίσουμε ότι δηλαδή το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεργαστούν είτε με ιδιωτικού φορεί ή με άλλου διεθνού φορεί σε αυτό το τομέα. Θα πρέπει λοιπόν να τονιστεί αυτή η ανάγκη. Επίση θα πρέπει να τονίσουμε και πάλι το ρόλο της γυναίκας ε, στο πλαίσιο των ειρηνευτικών μας ε, ε, αποστολών. Θα πρέπει δηλαδή να τονίσουμε και πάλι τις σωστές ε, διαστάσεις. Ε, και κάτι ακόμα το οποίο δεν μπορούμε να ξεχνούμε είναι η σημερινή άσκηση της πολιτικής από των Ηνωμένων Το αναφέρεται με πολύ ευγενικό τρόπο το ότι δηλαδή η εκλογή του Προέδρου Τραμπ ουσιαστικά μας κατέδειξε ότι δεν μπορούμε μέσα είναι βασιζόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει δηλαδή να τοποθετηθούμε τώρα με ε, σαφήνεια μόνοι μας και σε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Ε, θα κάνουμε πάντως κάποιες ε, προτάσεις για βελτιώσεις του κειμένου προκειμένου να καταστεί το σχέδιο της έκθεσης ακόμα καλύτερο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σκούζο Περμόη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι γνωστή η θέση της ΓΚΟΕ δεν αποδεχόμαστε την έκθεση αυτή. Ξέρετε το λόγο, επειδή θέλουμε διαφορετική ευρωπαϊκή άμυνα. Και κουλτούρα ειρήνης. Στην οποία δεν ταιριάζει μια επιθετική στρατηγική, ιδιαίτερα αυτή που βολεύει τις μεγάλες επιχειρήσεις όπλων. Ιδιαίτερα δεν θέλουμε να είμαστε υποτακτικοί του ΝΑΤΟ, μια, μιας αναχρονιστικής οργάνωσης. Υπό Αμερικανική διοίκηση, όπω ο τωρινός διοικητής. Νομίζω εδώ ακριβώς δείχνει πόσο υποτακτική είναι η Ένωση σε σχέση με το ΝΑΤΟ. Όπως είδαμε και σε όλες τις διασκέψεις κορυφής του ΝΑΤΟ άτομο το οποίο χρησιμοποιεί τις ε, δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα μέσα της ΠΕΣΚΟ. Εξάλλου ε, προτείνει, και το λέει επανειλημμένος, παπαγαλίγουστοντας, αυτά που λέει και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ για το στρατιωτικό σύγκελα, δηλαδή να μην υπάρχουν εμπόδια στις στρατιωτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην παρουσία του στην Ευρώπη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο εγώ είναι κατά και δεν θα στηρίξουμε την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπαλέρο. Ευχαριστώ. Δεν θα επισέλθω σε όλες τις λεπτομέρειες. Δεν θα σας πω ακριβώς και πλήρως την απόψή μας γιατί είναι γνωστή, αλλά να αναφερθώ σε κάποια επιμέρους ζητήματα του κειμένου. Διατύπωση. Ας πούμε εδώ που λέμε στο 8 για τις δυτικές αξίες νοικίες αξίες, τι είναι αυτό, τι περιλαμβάνει. Γιατί στο F μετά λέτε μέλη της Ανατολικής Ευρώπης, μέλη της Δυτικής Ευρώπης, τι ακριβώς εννοείται εδώ πέρα. Για την πιο ουσιώδη εταιρική σχέση πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν είμαστε όλοι χώρες ΝΑΤΟ, όπως η χώρα μας πούμε. Και δεν έχουμε τα ίδια στρατηγικά συμφέροντα. Οπότε μπορείτε να διευκρινίσετε σε ποιους αναφέρεστε. Γιατί τα στρατηγικά συμφέροντα δεν συμπίπτουν μεταξύ όλων των χωρών της Ένωσης. Δεν έχουμε τα ίδια συμφέροντα όλοι μας. Μετά ενίσχυση της εταιρικής σχέσης με το ΝΑΤΟ Διευκρινίστε μου, τι εννοείται εδώ. Μετά στο σημείο 5 έχουμε ένα ψήφισμα μετά τι επιθέσει στο Παρίσι ένα ψήφισμα στο 42-7 και ίσως αυτά που αναφέρονται εδώ να είναι κάπως αντιφατικά σε σχέση με αυτά που γράφαμε στο ψήφισμα. Ίσως θα πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό. Έχω και άλλα που θα μπορούσα να πω για να είμαι ακριβέστερη αλλά θα επανέλθω όταν θα συζητήσουμε τις τροπολογίες για τους ίδιους πόρους τώρα και στο, στο 9 και πιο κάτω στο 22 μιλάμε για τις χώρες που δεν είναι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και θα πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις τους προς το ΝΑΤΟ. Ποιες είναι αυτές οι υποχρεώσεις? Αφορά τι κάποιο ποσοστό σε σχέση με τις δαπάνες για αυτούς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Ναι, εντάξει, υπάρχουν εθελοντικές δεσμεύσεις, όχι όμως υποχρεωτικές. Γιατί εμείς συνεργαζόμαστε με το ΝΑΤΟ σε εθελοντική βάση. Στο 25 επίσης αναφέρεστε στην ανάγκη ενίσχυσης της τεχνολογικής και μηχανικής συνεργασίας μεταξύ ΝΑΤΟ και Ένωση. Ένωσης των χωρών μελών της βιομηχανικής βάσης. Όχι όμως της βιομηχανικής βάσης ως Ένωση ή ως ΝΑΤΟ. Μετά, η ναυτική διοίκηση του ΝΑΤΟ, η Frontex κλπ. Και η συνεργασία για τη μετανάστευση. Τι γίνεται εδώ. Έχουμε και άλλα σχόλια, αλλά αυτά προς το παρόν και θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Πάσκου, για την έκθεση αυτή, η οποία σίγουρα είναι μια καλή βάση κίνησης για τις μελλοντικέ συζητήσεις μας ε, και αναλύσεις. Προτού πάω στα πιο συγκεκριμένα, να θυμίσω το πλάσιο, το πλαίσιο στο οποίο κινούμεθα. Τα τελευταία χρόνια αλλάζει το παράδειγμα των σχέσεων αυτών, διότι αλλάζει το συνολικό πλαίσιο. Οι πολιτικές μπορούν να μετακινούνται, αλλά το πλαίσιο της ασφάλειας για την Ήπειρο την ευρωπαϊκή σήμερα είναι πολύ πιο συγκεκριμένο και πολύ πιο απαιτητικό από αυτό που ήταν πριν από κάποια χρόνια. Πρέπει να βλέπουμε λοιπόν και την εξωτερική δυναμική, τη σχέση την διατλαντική με τις Ηνωμένε Πολιτείες αλλά και την έρευνα που πρέπει να έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μια αυτονομία αμυντική. Βλέπουμε και στα πλαίσια της συζήτησης της δημοσιονομικής ότι δεν είναι πλέον ένα περιθωριακό ζήτημα και το βλέπουμε αυτό και στο Κοινοβούλιο. Πρέπει λοιπόν να διατηρούμε υπόψη ότι οι δύο οργανισμοί αυτοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, δεν είναι ταυτόσιμοι Στην έκθεση δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ε, αντιστοίχηση της, των αξιών που μοιράζονται οι δύο, το οποίο είναι σωστό αλλά πρέπει να διαρωτηθεί κανείς πώς τελικώς υλοποιείται αυτό. Στο σημείο 11 της έκθεσης για την ενίσχυση της συνεργασίας με το ΝΑΤΟ στην ανατορική διάσταση μου φαίνεται κάπως περιοριστική προσέγγιση όπως και στο τμήμα των ε, κυρίων σημείων συνεργασίας, μόνο στο σημείο 19 ε, αναφέρεται ένα μήνυμα αρκετά αποθαρρυντικό για τις ε, πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρούν ότι το ζήτημα της μετανάστευσης είναι άμεση απειλή για την Ευρώπη. Μία ενισχυμένη συνεργασία του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις, όλα τα σημαντικά θέματα πολιτικής και να είναι win-win για όλους και όχι να ευνοεί τη μία αντί για την άλλη πλευρά. Θα πρέπει να μην ξεχνούμε και τον άξονα Ανατολή Δύσεω και Βορρά Ανώτου, χωρί να ξεχνούμε τα Βαλκάνια και τα θέματα τη μετανάστευση. Κοινά σημεία είναι βεβαίω κοινέ ασκήσει, τυποποίηση των διαδικασιών, συνεργασία στην έρευνα τη βιομηχανική ε, ανάπτυξη αλλά η συνεργασία τελικώ τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ΝΑΤΟ θα πρέπει να βασίζεται σε κάποιου κοινού άξονε και όχι να απευθύνεται κατά τρίτων. Πρέπει λοιπόν να εξευρεθούν συνεργίες δομικέ που θα ανταποκρίνονται στι στις ε, των δύο πλευρών με τις ιδιαιτερότητε που διατηρούν. Ε, και βέβαια στο, κάτι που έχει ακόμα να εξετάσει κανείς είναι τις προθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια της νεασίας αυτής, αλλά ίσως αυτό θα μπορέσουμε να το εξετάσουμε στη μελλοντική συζήτηση που θα έχουμε για τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο μιλητής. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Βανόρντερ νομίζω ήθελε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώμη ε, που καθυστέρησα σήμερα αλλά δεν μπορούσα να βρίσκομαι στο ίδιο σημείο. Είχα πάρα πολλές υποχρεώσεις. Να ευχαριστήσω τον κύριο Πάσκου για το κείμενο που είναι εξαιρετικό, έχει πολλά θετικά σημεία και δεν είναι καθόλου έκπληξη που μας υποβάλλεται ένα απολύτως ισορροπημένο κείμενο σε σχέση με την ε, συμμαχία με τον ΑΤΟ. Έχουμε κάποιες προτάσει τροπολογιών, αλλά όπως γνωρίζετε, Πρόεδρε, έχουμε ένα κύριο πρόβλημα με το βασικό άξονα του USDP ε, και της Ευρωακής Αμυντικής μηχανίας και επανέρχομαι στο γνωστό ρητό της κυρίας Όλμπραιτ, μετά τη συνέντευξη ΛΟ, για τα 3D dealing, discrimination και είναι ακόμα σχετικά αυτά σήμερα συνάδελφε. Γιατί δεν ξέρουμε πώς θα αναπτυχθεί το ΠΕΣΚΟ. Ήδη η γαλλική ε, σκέψη ότι θα πρέπει να συνεργαστούν οι πιο ικανοί και πιο ισχυροί έχει ξεπεραστεί γιατί όλοι συμμετείχαν στο ΠΕΣΚΟ. Επομένω, καθόλου δεν καταλαβαίνουμε τι είναι το ΠΕΣΚΟ, ποια είναι η φιλοδοξία. Ακούς, ακούμε όρους όπως στρατηγική αυτονομία, αλλά κανείς δεν τους έχει ορίσει. Γιατί προσπαθώντας να τους ορίσει κανείς, θα φτάναμε σε σοβαρές αντιφάσεις. Και δεν μιλώ για το δικό μου κράτος μέλος, μιλώ για τα υπόλοιπα 27. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα θεμελιώδεις δυσκολίες και έχω την εντύπωση ότι δημιουργούμε εδώ ένα οικοδόμημα και μιλούμε για τη σχέση μας με τον ΝΑΤΟ την ώρα που βεβαίως τα περισσότερα κράτη-μέλη είναι μέλη του ΝΑΤΟ, λέει ο μιλητής. Ο Σουηδός ε, συνάδελφος λέει ότι δεν, υπάρχουν, ότι δεν είναι ακριβώς με ε, τα στρατηγικά συμφέροντα. Ε, είναι όμως, θα έλεγα εγώ η Σουηδία και η Φιλανδία είναι δύο από τους καλύτερους συμμάχους του ΝΑΤΟ και αν ε, προέκυπτε η ανάγκη ε, από το ΝΑΤΟ θα εξαρτώσασταν για την άμυνά σας. Ε, το γνωρίζουμε όλοι, αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε. Λέει ο Μίλτης. η Εβραϊκή Συνθήκη γράφει για την αμυντική βιομηχανία μαζί με μια ρήτρα διαφυγής βεβαίως σχετικά με τον Άτο και τις ε, ευθύνες που αναλαμβάνουν ε, τα κράτη-μέλη. Εν πάση όλο αυτό το εγχείρημα κινείται σε μια λανθασμένη κατεύθυνση, ε, πιστεύω, αλλά η έκθεση καθεαυτή είναι αρκετά ισορροπημένη, θα υποβάλουμε τα σχόλιά μας εγκαίρως. Σας ευχαριστώ, η κυρία Κλέρ Μούντι έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε χρόνια για αυτήν την εξαιρετική έκθεση. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα-δύο σημεία από την πλευρά μου. Το ένα από αυτά είναι την οποία έθεσε ο συνάδελφος Τενταζόν και άλλοι σε ό,τι αφορά τη διάκριση που θα πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στις δύο, στους δύο οργανισμούς, τις διαφορές δηλαδή μεταξύ τους και το γεγονός ότι θα πρέπει να αναγνωρίζουμε αυτές οι διαφορές. Συμφωνώ με αυτό. Ε, και λίγο α, παρεκκλίνω από αυτό που είπατε συνάδελφε σε ό,τι αφορά αυτή τη διαφοροποίηση σε σχέση με την άμυνα στον κυβερνοχώρο. Δηλαδή, ε, αυτές οι διαφορετικές αφετηρίες αν θέλετε, ε, δηλαδή η πολιτική αφενός, η μη στρατιωτική και η στρατιωτική αφετέρου, ουσιαστικά ε, συνενώνονται εδώ σε ό,τι αφορά τον ε, κυβερνοχώρο και πραγματικά η διαφορετικότητα των δύο οργανώσεων έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα, δηλαδή μπορούν ε, να καταστούν ακόμα ισχυρότερε ε, στο πλαίσιο της συνεργασία τους παρέχοντας περισσότερη προστασία στους πολίτες μας. Από εκεί και μετά αυτό που είπατε ότι δεν θα πρέπει ε, απλώς να συνεργάζονται οι οργανισμοί μεταξύ τους, αλλά να γίνεται και αυτό ορατό προς τα έξω. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικότερα στη σημερινή χρονική συγκυρία, δηλαδή το ζήτημα της επικοινωνίας, της ε, προβολής αυτής της συνεργασίας προς τα έξω. Ε, δύο ακόμα σχόλια θα ήθελα να κάνω. Είναι καταρχήν σε ό,τι αφορά την, την συντονισμένη αξιολόγηση ε, και τον τρόπο που γίνεται ο υπολογισμό των δαπανών. Προφανώ λαμβάνουμε υπόψη μα το διαφορετικό χαρακτήρα των δύο οργανώσεων, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την ανάλυση των κοινών η οποία θα πρέπει να γίνει και ε, ε, κατά συνέπεια τον συντονισμό που θα πρέπει να λάβει η χώρα. Και δεύτερο, σε ό,τι αφορά το συντονισμό και αυτόν τον στόχο του ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά το, την δαπάνη του προπολισμού κατά 20% σε ε, δραστηριότητε ε, έρευνα και ανάπτυξη. Ναι, προφανώ θα πρέπει να παραμείνει αυτό ο στόχο. αλλά σε ό,τι αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη, αν υπάρχει απόκληση ό,τι αφορά του στόχου μας, τότε αυτή θα πρέπει να υπάρχει συνειδητά. Δηλαδή, συνειδητά θα πρέπει να επενδύουμε σε διαφορετικού είδου μέτρα σε αυτέ τι περιπτώσει. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Ε, κύριε Πάσκο, έχετε για μία ακόμα φορά το λόγο. Α, όχι πολύ σύντομα να πω και εγώ ότι πρόκειται για μια πολύ ισορροπημένη έκθεση. Θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι το οποίο αναφέραμε και στο πλαίσιο τη συζήτηση που κάναμε σήμερα το πρωί σε ό,τι αφορά την άμυνα στον κυβερνοχώρο, ότι δηλαδή θα πρέπει να δημιουργήσουμε και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα περισσότερε ικανότητε σε ό,τι αφορά την κυβερνοάμυνα όπως ανέφεραν δηλαδή και άλλοι συνάδελφοι, θα πρέπει να προβλέψουμε τις εργασίες που θα κάνουμε στο μέλλον ε, ώστε να είμαστε πιο συντονισμένοι και προκειμένου να χαρτογραφήσουμε το εισαγωγικό της ανάγκης ε, των διαφορετικών κρατών μελών, αφού δεν έχουμε ακόμα κατανέμει τι ε, αρμοδιότητε μεταξύ μας. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρε, ο κύριος Πασκού. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για αυτές τις προτάσει. Γνωρίζω ότι πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία δεν είναι κάτι το οποίο έχει καταλήξει αυτής εξ αρχής. Ούτε αυτός είναι ο στόχος μου. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για τα ίδια ζητήματα. Και αυτό ίσως να σημαίνει ε, υπερβολικά συχνά. Αλλά σε κάθε περίπτωση αναμένουμε ενδιαφέρον τις τροπολογίες σας, αν θα τις εξετάσω. Ε, με γνωρίζετε ούτως ή άλλως, έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν, οπότε εγώ δεν έχω έτσι ε, προδεκάσει το πώς θα διαμορφωθεί το τελικό κείμενο. Έχω κάποια ατζέντα. Πάντως, εάν το ΝΑΤΟ αποτελεί πραγματικά την έκφραση της διατλαντικής συμμαχίας, γιατί όλοι θέλουμε να είμαστε ασφαλείς απέναντι στη ρωσική απειλή, τότε ναι, γνωρίζουμε πως όλοι θέλουμε να συνεργαστούμε γιατί όλοι θέλουμε να είμαστε ασφαλείς απέναντι σε αυτή τη ρωσική απειλή. Και το ΝΑΤΟ μέχρι στιγμής αποτελούσε την έκφραση αυτής της υπερατλαντικής συμμαχίας. Σε ό,τι αφορά όμως την Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύει το ότι πρόκειται για την έκφραση της υπερατλαντικής, του υπερατλαντικού ανταγωνισμού, αμπορικού ανταγωνισμού και άλλων. Άρα λοιπόν αυτή η προσπάθεια, η έναρξη της προσπάθειας που έγινε σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Άμυνα ξεκίνησε αν θέλετε από αυτό το σκεπτικό του ανταγωνισμού έναντι των ε, ΗΠΑ. Πάντως, ε, Αρνό, έχεις δίκιο σε αυτό που είπε, ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε λίγο περισσότερο ε, την διάσταση της διαφορετικότητας μεταξύ των δύο διαφορετικών οργανισμών, παρότι αυτοί συνεργάζονται. Το πρόβλημά μου είναι ότι μόλις ε, εισέλθει στο αμυντικό τομέα Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν αποτελεί ε, αμυντικό οργανισμό, τότε θα πρέπει να υιοθετήσει τους ίδιους κανόνες παιχνιδιού με αυτούς που εφαρμόζει το ΝΑΤΟ. Και τίθεται εδώ το ερώτημα, μπορούμε πράγματι να ε, εφαρμόσουμε διαφορετικούς κανόνες, για παράδειγμα, ή θα πρέπει να ακολουθήσουμε τους ίδιους κανόνες με αυτούς που χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ. έχω κάποιες αμφιβολίες δηλαδή ως προς το πώς θα το επιδείχουμε αυτό. Αλλά όπως είπατε και εσείς, οι δύο αυτοί οι οργανισμοί θα πρέπει να αναγνωρίζουν τις διαφορές τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Βερολίνο Plus, το Berlin Plus, υπήρξε μία απόπειρα εξέβρεσης πρακτικών λύσεων, λαμβάνοντας υπόψη το ότι και οι δύο αυτοί οι οργανισμοί δραστηριοποιούνται στον χώρο της ε, διαχείρισης κρίσεων παρά τις διαφορές τους. Υπήρξε λοιπόν η πρόταση μια σειρά εργαλείων τότε και γι' αυτό το ΝΑΤΟ έχει σε αυτό το πλαίσιο την προτεραιότητα. Δηλαδή εκείνο θα πρέπει να πει αν θέλει να αξιοποιήσει όχι αυτά τα εργαλεία και αν δεν επιθυμεί στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνει. Το ΝΑΤΟ ήδη ανέφερε ότι θέλει να συμπεριλάβει και μία μη στρατιωτική διάσταση σε αυτή την εργαλειοθήκη Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω το, η μεγάλη δοκιμή, το τεστ θα είναι ε, η συμμετοχή του ΝΑΤΟ σε μία ε, επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι αλλού. Αλλά λοιπόν εδώ πώς το ζητούμενο είναι να επιτύχουμε την αύξηση της προστασίας των πολιτών μας στο πλαίσιο μιας τέτοιου είδους συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών οργανισμών. Αυτό έχω κατά νου. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση νομίζω πως το Βερολίνο Plus ενδεχομένως θα πρέπει να προσαρμοστεί. Δεν ξέρω βέβαια αν θα παραμείνει το ίδιο ή αν θα βελτιωθεί ή βέβαια το αντίθετο αν θα επιδεινωθεί. Πάντως νομίζω πως έχει φτάσει η χρονική στιγμή να εξετάσουμε τη δυνατότητα τέτοια συνεργασία όχι μόνο σε ό,τι αφορά την ε, διαχείριση κρίσεων, αλλά και σε σχέση με άλλου τομεί. Σε ό,τι αφορά αυτό που επιτερήσει. Ναι, υπάρχει διαφορετική στρατηγική οπτική γωνία σε ό,τι αφορά τις Ανατολικέ χώρες και τις δυτικές ε, χώρες. Ε, σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τη Ρωσία, οι δυτικές ε, χώρες ε, την ε, θεωρούν ως ε, λιγότερο απειλητική από ό,τι ανατολικές χώρες και θεωρούν μάλιστα πως είναι, μπορεί να αποτελέσει και μια ευκαιρία επιχειρηματική. Αλλά οι ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες έχουν μια ιστορία με τη Ρωσία, ένα ιστορικό και γι' αυτό την αντιμετωπίζουν κατά κύριο λόγο ως γεωπολιτικό παράγοντα και όχι ως εμπορικό εταίρο. Αυτό είναι αυτό που ισχύει τη σήμερα ημέρα. Αλλά όπως είπε ο Τζόφρεϊ, δεν νομίζω πως η Σουηδία ή η Φιλανδία εφαρμόζουν τελικά ή έχουν διαφορετικά στρατηγικά συμφέροντα από τους υπόλοιπους. Και αυτό ίσχυε και κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Δηλαδή το ΝΑΤΟ ε, ε, ήταν εκείνο που έγινε την ασφάλεια και της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Δεν ήταν άλλη οργάνωση η οποία εγγυόταν την ασφάλειά τους. Και όπως είπαμε είναι πολύ καλή συνεργασία με το ΝΑΤΟ που έχουμε αυτή τη στιγμή και κανένας δεν την επιβάλλει σε μας. Απλώς αυτό που είπα ότι θα πρέπει να μεταχειριζόμαστε ισότιμα τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ε, χρήζουν ε, τη ίδια προστασία οι πολίτε του με του πολίτε των 100 μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα το καταστήσω αυτό σαφέστερο στο κείμενό μου, αν αυτό χρειάζεται. Κύριε Καστάντου, όταν αναφέρθηκα στο Βορρά και το Νότο, ε, αναφερόμουν σε ζητήματα μεταφορών. Τίποτα άλλο. Ε, όχι δηλαδή στην ε, οικονομική ή ε, αυτή η άλλη διάσταση. Απλώς είπα ότι από τότε που διαλύθηκαν τα μεγάλα στρατεύματα του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη, υπόθηκε ότι θα πρέπει να είναι δυνατή η επιστροφή εκεί, η επαναδραστηριοποίηση, αφήνοντας μικρότερα τμήματα. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άξονες μεταφοράς που είχαν δημιουργηθεί, όλοι αυτοί οι διάδρομοι, αφορούσαν ακριβώς αυτές τις δυνατότητες ε, μεταφοράς από στρατιωτικής άποψης και μεταξύ Βορρά και Νότου. Και άρα λοιπόν η αναφορά που έγινε σε Βορρά και Νότου έγινε σε αυτό το πλαίσιο και μόνο. νομίζω πως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Ορισμένους σε φόβους, ότι αν αναθέσουμε πάρα πολλά σε, ένα, στον ένα στον άλλο οργανισμό ενδεχομένως θα ε, είναι υπερβολικό. Νομίζω πως τα όσα αφορούν τα αμυντικά ζητήματα του ΝΑΤΟ θα πρέπει να παραμένουν ακριβώς στις χώρες ε, μέλη του ΝΑΤΟ. Και γι' αυτό θα πρέπει να δείξουμε λίγη περισσότερη εμπιστοσύνη σε αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω πως γνωρίζετε όλοι σας ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν αυτές οι διαφορές, θα συνεχιστεί η ενίσχυση της συνεργασίας και ελπίζω πως η νέα διακήρυξη που θα γίνει σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα αποτελέσει μια συνεισφορά για περισσότερη δηλαδή συνεργασία, περισσότερα στοιχεία συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών και όχι λιγότερα. Και δεν θα πρέπει να μα αποθαρρύνει το γεγονό ότι δεν ε, πετύχαμε πολλά σε ό,τι αφορά δηλαδή τη συμπερίληψη στοιχείων στην πρώτη διακήρυξη. Και νομίζω πως ακόμα βρισκόμαστε σε μια φάση εκόλαψης αν θέλετε αυτής της ενίσχυσης της συνεργασίας προετοιμασίας σε μια προκατακτική φάση. Αυτά από την πλευρά μου σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Συνάδελφοι, να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι 28 Μαρτίου. Για τη δεύτερη εξέταση της έκθεσης και των τροπολογιών είναι η 15 Μαΐου και μετά θα ψηφίσουμε στην ΑΦΕΤ την επόμενη, 16-17 Μαΐου. αν θέλουμε να τελειώσουμε στο εξάμεινο και να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια τον Ιούνιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παραμείνετε εδώ, γιατί το επόμενο σημείο στην ημερήσια είναι ενημέρωση για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 6ης Μαρτίου. Ανταλλαγή απόψεων με τον Πέδρο Σεράνο, αναπληρωτή γενικό γραμματέα της ΕΕΔ. Colleagues, once more, Ενημέρωση για το Συμβούλιο Εξωτερικών Προθέσεων Άμυνας. Ο προσδευτής Πέδρος Εράνου θα μας ενημερώσει, ο οποίος συχνά πρόσφατα μας ενημερώνει για σημαντικά συμβάντα. Καλώς ορίσατε, κύριε Πρεσβευτά. Λυπόμαστε για την καθυστέρηση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Με χαρά σας ξαναβλέπω. Είδα ότι είχατε συζήτηση για τις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ένωσης. Δεν ξέρω αν χρειαστεί να πω κάτι ιδιαίτερο. Όχι, πείτε ότι γουστάρετε, λέει η Πρόεδρος. Μου παν, πάντως θα πρέπει να σας ενημερώσω και θα μιλήσω έτσι γενικά. Πρόεδρος, συζητήσαμε την έκθεση του κύριου Πάσκου για πρώτη φορά, αυτή την έκθεση πρωτοβουλία. Ωραία λέει ο να σα ενημερώσω εγώ. Συμβούλιο λοιπόν Άμυνα. Να σας ενημερώσω. Καταρχάς, εκτιμούμε τη δουλειά της Επιτροπής σας και ακούμε με πολύ προσοχή τις υποδείξεις και τις παρατηρήσεις σας. Έκτη Μαρτίου λοιπόν έγινε αυτό το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων Άμυνας. Συζητήθηκε το θέμα της μόνιμης ε, δομής συνεργασίας ΠΕΣΚΟ. Πρώτη φορά που υιοθετεί αποφάσεις στο Συμβούλιο στο πλαίσιο ΠΕΣΚΟ όλες οι χώρες που ήταν παρούσες συμμετείχαν σε αυτή την επίσημη λήψη αποφάσεων σχέση με κάποια προγράμματα και είχαμε μια σύσταση το οποίο είναι το άλλο νομικό μέσο που διαθέτει το Συμβούλιο στα πλαίσια της, του σχήματος ΠΕΣΚΟ είναι ένας οδικός χάρτης για την εφαρμογή της ίδιας της ΠΕΣΚΟ αλλά βέβαια και η συζήτηση πήγε παραπέρα ήταν μια συζήτηση που αφορούσε την γενική στρατηγική για τα θέματα άμενας και ένα follow-up σε σχέση πάντα με την ΠΕΣΚΟ. Μετά είχαμε τα λόγια απόψεων για τις σχέσεις ΕΕΝΑΤΟΥ, κατά το παρουσιακό πια σε συναντήσεις Συμβουλίου, Εξωτερικών Θέματα Άμυνας όπου συμμετέχουμε και ένα το θέμα στη μέση διάταξη που συζητήσαμε ήταν οι μη εκτελεστικές στρατηγικές αποστολές Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή εκπαιδευτικές αποστολές Σομαλία, στο Μαλί κλπ. Για θέματα τώρα ασφάλειας και άμυνας κοιτάξαμε, τα κυριότερα θέματα προτεραιότητας για φέτος. Κύρια διαπίστωση από όλου τους υπουργούς ήταν ότι αυτό που είναι σημαντικό τώρα είναι να εφαρμόσουμε όλες αυτές τις προτεραιότητες που έχουν ξεκινήσει ώστε να παράξουμε κάποια αποτελέσματα και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό ιδιαίτερα στο πακέτο που αφορά την εξέλιξη ε, ικανότητας για την άμυνα. Εδώ έχουμε να κάνουμε το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο, με την ΠΕΣΚΟ, κάτι στο οποίο βεβαίω θα συμμετέχετε κι εσείς αν δεν συμμετέχετε ιδιαίτερα στο EDITP και επίσης συζητήσαμε για το πώς ακριβώς θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτό το πακέτο με τρόπο συνεκτικό. Αν δούμε τις διάφορες τροπολογίες δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εδώ προέχει αυτή η δυνατότητα ανάπτυξης αμυντικών ικανοτήτων. Θα έχουμε το καλοκαίρι μια αναθεώρηση για να δούμε πού βρισκόμαστε και αυτό επίσης θα συνοδευτεί με την ετήσια αναθεώρηση για θέματα άμυνας, όπου ξέρετε ότι είναι κάτι αυτό που κάνουν ετησίως οι χώρες μέλη, ώστε να εντοπίσουμε ακριβώς τα κενά στο στρατιωτικό σκέλος και μετά έχουμε την μόνιμη ειδοποίηση εργασία στην ΠΕΣΚΟ, όπου εκεί συμβάλλουν όλες οι χώρες για την αντιμετώπιση και εκπλήρωση αυτών των προκλήσεων. σε συνεργασία πάντοτε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα και το EDIDP για να δούμε ακριβώ πώς προχωράει όλη η διαδικασία. Για να δούμε ακριβώ πώς θα έχουμε προγράμματα τα οποία θα οδηγήσουν σε μια ουσιώδη ανάπτυξη αμυντικού δυναμικού. Συζητήσαμε με την Κομισιόν και με συναδέλφους για το ποιοι θα ήταν οι κατάλληλοι μηχανισμοί ώστε να έχουμε τη σωστή αλληλουχία στον εντοπισμό αυτών των προγραμμάτων και των διαδικασιών αξιολόγησης. Αυτό λοιπόν το συζητήσαμε με τους υπουργούς, υπήρξε ευρεία συνένεση γι' αυτό. Άλλο ένα ζήτημα, το οποίο συζητήθηκε ευρέως, ήταν η στρατιωτική κινητικότητα. Έχει να κάνει με το σημαντικό θέμα της συνεργασία μας με το ΝΑΤΟ έχει να κάνει και με το EDIDP. Στρατιωτική λοιπόν κινητικότητα, τι μπορεί να κάνει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει τις χώρες μέλη ώστε να διασφαλίσει μια ταχεία μετακίνηση υλικού και δυνάμεων στην Ευρώπη και όπου άλλο χρειάζεται. Εδώ έχουμε να κάνουμε με διπλωματικές δηλαδή ρυθμίσεις, ε, θέματα πρακτικά, θέματα υποδομής, μαζί με ένα σχέδιο δράσης που θα υποβληθεί από την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο τώρα στο τέλος του μήνα, όπου να είναι δηλαδή. Και το τελευταίο θέμα που ζητήσαμε εδώ ήταν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Ειρήνης. Ένας μηχανισμός δηλαδή που χρηματοδοτείται εκτός προπολογισμού που χρηματοδοτείται βεβαίως από τον προπολογισμό για τις στρατικές επιχειρήσεις αλλά και από τα κονδύλια που αφορούν τις εταιρικές μας σχέσεις ας πούμε για παρεμβάσεις στην Αφρική. Εκεί εξετάσαμε το πώς ακριβώς θα μπορούσαμε να δώσουμε υποστήριξη σε εξοπλισμό των εταίρων, αυτό που ονομάσαμε CBST μετά την ε, αναθεώρηση που έγινε. Εμείς έχουμε περιορισμού στον προπολογισμό. Κοιτάξτε λοιπόν πώς θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε αυτούς τους ε, δημοσιονομικού περιορισμού για να χρηματοδοτήσουμε αυτή την νέα δομή. Αυτό λοιπόν συζητήσαμε σε επίπεδο υπουργών και οι υπουργοί με ενδιαφέροντα συζήτησαν όλα αυτά. Τώρα για το ΝΑΤΟ. Ο αρχηγός του ΝΑΤΟ δεν ήρθε. Εκπροσωπήθηκε από τον ε, κύριο Γκέτε Μίλλερ τον βοηθό του. Κοιτάξαμε λοιπόν το πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στις αμοιβέ μας σχέσεις. Ήδη έχουμε αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλειών, 74 δηλαδή δράσεις τις οποίες έχουμε εντοπίσει και από αυτές τις δράσεις οι περισσότερες δεν θα ολοκληρωθούν με την εφαρμογή, αλλά ήδη αποτελούν μια διαδικασία συμμετοχής συνεχόμενη σε, αυτές τις, σε αυτούς 7 τομείς που έχουμε εντοπίσει με τις αντίστοιχε δράσεις, αλλά εδώ ακριβώς εμπλέκουμε τις διάφορες οργανώσεις μας για να συνεργαστούν στα πλαίσια αυτών των 7 τομέων που γνωρίζουμε, δηλαδή επιχειρήσεις, ανάπτυξη δυναμικού, κυβερνοχώρος, τα βιομηχανία, η και συνεργασία με τους εταίρους μας. Μια μακροσκελής δηλαδή λίστα, όπως βλέπετε. Και θα ήθελα τώρα να αποφερθώ σε ευκαιρίες για να διευκρινίσω, επειδή ακριβώς υπήρξαν κάποιες ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με το ότι τα τελευταία χρόνια αυτά που κάναμε στην Ένωση για να προωθήσουμε πρωτοβουλίες άμυνας ήταν ευπρόσδεκτα, αλλά ιδιαίτερα από το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, αλλά υπήρξαν κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με την υποστήριξη δράσεων του ΝΑΤΟ. Και εδώ ήταν χρήσιμη από αυτού η συνάντηση για να τονίσουμε ακριβώς το ότι αυτά που κάνουμε στην Ένωση θα ενισχύσουν και το ΝΑΤΟ το ότι αυτές οι νέες δράσεις αφορούν κυρίως τη δυνατότητα χωρών μελών και βεβαίως είναι δυναμικό που χρησιμοποιείται και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και υπάρχει σωστή συνεργασία μεταξύ προσωπικού. Τονίστηκε επίσης το θέμα της κινητικότητας και των προγραμμάτων κινητικότητας που διαθέτει αυτή τη στιγμή πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση και που βοηθά τον ΝΑΤΟ να ξεπεράσει δυσκολίες. Το οποίο όμως ε, θα ήταν δύσκολο να γίνει εκτός πλαισίου Ένωσης η ΝΑΤΟ. Πρέπει να δούμε λοιπόν εδώ τι γίνεται με τις υποδομές σε περιπτώσει όπου το ΝΑΤΟ δεν έχει δυνατότητα κινητοποίησης από μόνο του. Εμπλέξαμε και το ΝΑΤΟ από την αρχή σε αυτές τις διαδικασίες όπως ξέρετε. Ξεκίνησαμε μια ομάδα εργασίας υπό το EDA παρήγαγε αυτή η ομάδα ένα οδικό χάρτη και κάποιοι από τους συνοδικού συμμάχους ήδη συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα εργασία και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με αυτού, όσο προχωράμε με το σχέδιο δράσης το οποίο έχει προβλεφθεί. Αυτό το τόνισαν λοιπόν όλοι και εκτιμήθηκε από τον βοηθό του Γενικού Γραμματέα. Αυτό λοιπόν ως όλη η δικασία διευκρίνησε κάποια πράγματα, διασκέδασε κάποιες ανησυχίες και το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να θίξω αφορά την Πέσκο από την Σκοπιά της Συνεργασίας. Είπα νωρίτερα ότι είχαμε δύο κύριες αποφάσεις που λήφθηκαν. Μια απόφαση για τα ίδια τα προγράμματα της ΠΕΣΚΟ που είχαν ανακοινωθεί το Δεκέμβριο όταν είχε θεσπιστεί η ΠΕΣΚΟ και ο δικός χάρτης για την ίδια την εφαρμογή της ΠΕΣΚΟ. Και οι υπουργοί συμφώνησαν να συνεχίσουμε την προσπάθεια και να δοθεί όθεση ώστε να πετύχουμε αποτελέσματα. Επίσης, συμφώνησαν για τα άμεσα τρία βήματα μέχρι τον Ιούνιο που θα πρέπει να γίνουν, δηλαδή η απόφαση που θα παρουσιαστεί τον Ιούνιο σε σχέση με την κυβέρνηση των προγραμμάτων, Δεύτερον, η συμφωνία σε σχέση με την αλληλουχία της εφαρμογής των δεσμεύσεων στα πλαίσια της ΠΕΣΚΟ και τρίτον, η έναρξη, η κίνηση μάλλον μιας νέας δέσμης προγραμμάτων που θα πρέπει να ξεκινήσουν πριν το καλοκαίρι. όπω επίση και τέταρτο σημείο η συμμετοχή των χωρών στην ΠΕΣΚΟ. Και υπάρχει επίση, όπω ξέρετε, και συμφωνία να τα εξετάσουμε όλα αυτά πριν το τέλο του χρόνου. Υπήρξε λοιπόν εδώ συμφωνία και ομοφωνή σε σχέση με το να προχωρήσουμε για τα πράγματα τη ΠΕΣΚΟ. Και τελευταίο σημείο, και εδώ θα σταματήσω, είχαμε συζήτηση για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, τις μη εκτελεστικές, κεντρική Αφρική, Σομαλία, Μαλή κτλ. Αποστολές οι οποίες αφορούν κύριες στρατηγικές περιοχές για τα συμφέροντα της Ένωσης, αυτό που ονομάζουμε ζώνη ασφαλείας και αφορά την ασφάλεια της περιοχή, της περιοχής, τους βόρους και νοτιούς γείτονες της περιοχής, αλλά και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος, της τρομοκρατίας και αυτές οι επιχειρήσεις ε, είναι εμπροστοβαρής και σε σχέση με το Σαχέλ και αφορούν ιδιαίτερα αυτέ τι πέντε χώρες της ε, περιοχής και την υποστήριξή τους ιδιαίτερα για τη Σομαλία, ε, για την υποστήριξη της ε, μετάβασης προς τις ένοπλες δυνάμεις τη Σομαλίας. Η είπατε εκπρόσωπος τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη επάνδρωση αυτών των επιχειρήσεων, δηλαδή οι χωρισμοί θα πρέπει να συμβάλλουν με του απαραίτητου πόρου και υπήρξε θετική ανταπόκριση από πολλού υπουργού για το θέμα αυτό σχετικά, όπω επίση και για την επάνδρωση του στρατιωτικού σχεδιασμού όπου είχαμε κάποια κενά. Αυτά σε σχέση με την συνάντηση του Συμβουλίου για τα θέματα άμενας. Ξεκίνησαμε καλά για το τρέχον έτος, έτος που θα είναι που θα χαρακτηρίζεται από μια κύρια λέξη, δηλαδή εφαρμογή implementation. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά τον πρέσβη. Δεν ξέρω, η συνάδελφη, ο κύριος Ντανζό, θα ήθελε κάποιος να σχολιάσει. Sorry, Mrs. Valero. Η κυρία Βαλέρ. Ναι, μια πολύ σύντομη ερώτηση. Αναφερθήκατε ένα, για ένα εναλλακτικό του CPSD εκτός του ISP. Γιατί είχαμε προτείνει και την ε, τροποποίηση του Αθήνα ε, ακριβώς γι' αυτό. Αν μπορείτε λίγα περισσότερα να μας πείτε. Okay. Please. Ζητώ συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος. Δεν θέλω να σας εξωθήσω να μιλήσετε. Ο κύριος Βανάρντεν. Ναι, είμαι συνήθως έτσι επιφυλακτικός, Πρόεδρε, φοβούμαι ε, μήπως συζητήσατε τις, ε, τον αντίκτυπο επί των αμυντικών θεμάτων του Brexit. Ε, ήταν ε, θέμα που συζητήθηκε καθόλου αυτό και μια ερώτηση που δεν έχει σχέση με την 6η Μαρτίου. Τι άποψη έχει η, η ΕΔ επί της επιστολής του Πρόεδρου Γιούνκερ προς τον Πρόεδρο Πούτιν την οποία ε, κάποιοι θεωρούν απολύτως απαράδεκτη επί τη βάση των όσων έλαβαν χώρα ε, με την χημική επίθεση της Ρωσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο λέγει ο ομιλητής. Διερωτώ λοιπόν κατά πόσον και αυτό συζητήθηκε στην ΕΕΔ. Um, I ε, Και εγώ να προσθέσω μια ερώτηση. Ε, κυρία Σεράνο, αναφερθήκατε στο Συμβούλιο Πέσκο. Είναι κάτι το οποίο έχει μπει σε μια διαδικασία επισημοποίησης. Ε, αυτό ή απλώς μιλούμε για χώρες που συμμετέχουν και συναντώνται σε ένα κάποιο πλαίσιο. Ο κύριος Φρουζουλίκα, ευχαριστώ πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα σε σχέση με μια γνωμοδότηση της ΙΕΔ για την ρήτρια 42 της συνθήκης σε σχέση με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και δεδομένου του ότι ήδη την επικαλέστηκε η Γαλλία το 2015 και τώρα ε, συζητούμε ότι ίσως και το Ηνωμένο Βασίλειο να την επικαλεστεί κυρίως με τον ΝΕΤΟ, με τον ΝΑΤΟ αλλά ίσως και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΒ τι θεωρεί ότι αυτή η ρήτρα για την άμυνα, την αμοιβαία άμυνα θα πρέπει να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα γιατί αναφέρεται μόνο σε στρα... ανάληψη στρατιωτικής δράσης κατά κράτους μέλους χωρίς να αναφέρεται στις απειλές του κυβερνοχώρου που συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο 5, υβριδικές και τα λοιπά πρόσφατη της πρόσφατης επίθεσης στο Ηνωμένο Βασίλειο που θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει χημική επίθεση σε έδαφος κράτους μέλους. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι ο κύριος Πρέσβης τώρα μπορεί να απαντήσει σε αυτά και ίσως να μπορέσουμε να μας επιτρέψει ο χρόνος να έχουμε και ένα μικρό δεύτερο γύρο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε για το 42-7 σε σχέση με το 5. Αυτά τα άρθρα είναι, οι διατάξει αυτές είναι διαφορετικής φύσεως. Ο ρόλος του άρθρου 5, η συλλογική άμυνα ε, και τα αποτρεπτικά μέτρα και ο αποτρεπτικός χαρακτήρας του ΝΑΤΟ όλα αυτά αναγνωρίζονται ρητά από τη συνθήκη. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια ασυμβατότητα. Το άρθρο 42.7 είναι μια πολύ ευέλικτη διάξη. Αναφέρεται σε στήριξη κρατών μελών και όχι ενωσιακών δομών και αναφέρει ένα καθήκον αλληλεγγύης. Το επικαλέστηκε η Γαλλία μόνο μία φορά υπό δραματικότατες συνθήκες και τότε η Γαλλία είχε αποφασίσει ότι θα συζητήσει επιμέρους από κάθε κράτος μέλος πώς θα μπορούσε να βοηθήσει. Πρόκειται λοιπόν για μια διάταξη όπως σας έλεγα πολύ ευέλικτη. Δεν νομίζω ότι σε καμία περίπτωση έρχεται σε αντίφαση με τις ε, διατάξεις του άρθρου 5 που αφορούν τον ΝΑΤΟ. Μάλλον του ΝΑΤΟ. Είναι όμως ένα σημαντικό στοιχείο αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα για τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Και σε αντίθεση με το 222 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει πολύ σαφείς διαδικασίες για το πώς θα υλοποιηθεί, ιδιαίτερα μέσω του ICPR. Εδώ δεν έχουμε διαδικασίες είναι η ίδια, το ίδιο το κράτος μέλος που επικαλείται τη διάταξη προκειμένου να ζητήσει αλληλεγγύα από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη με τα μέσα που έχουν τους. Και όταν επικλήθηκε από τη Γαλλία, παρότι δεν αναφερόταν τα συνθήκη, είχαμε αναφερθεί στη δυνατότητα ε, συνεπικουρία των οραϊκών δομών. Εν πάση υπάρχει ευελιξία. Και είναι πολύ διαφορετικό από το άρθρο 5 του Βορειοατλαντικού Ατλαντικού Συμφώνου. Και δεν υπάρχει καμία συμβατότητα παραλαμβάνω. Τώρα, για τη δομή ΠΕΣΚΟ, όλοι λέμε ΠΕΣΚΟ format, οι νομικές μας υπηρεσίες βεβαίως μας συνιστούν να μην χρησιμοποιούμε την ορολογία ΠΕΣΚΟ format. Το Συμβούλιο είναι το Συμβούλιο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με τους κανόνες της ΠΕΣΚΟ που περιγράφονται από τη συνθήκη, δηλαδή μόνο τα συμμετέχοντα κράτη συμμετέχουν και στη διαδικασία λήψης απόφασης. Ενώ όλα τα κράτη-μέλη μπορούν να είναι απαρόντα και να παρεμβαίνουν και το έχουν πράξει κατά τη διάρκεια συζήτηση τέτοιων θεμάτων. Όμω, έχετε δίκιο, δεν ξέρω αν χρησιμοποίησα αυτή, αυτά τα λόγια, αυτή την ορολογία, Πρόεδρε, αν το έκανα έσφαλα. Αλλά το έχουμε κάπως συνηθίσει. Γιατί δίδει μια εικόνα, όμως ε, νομικός μιλώντας είναι, δεν είναι η ορθή ορολογία. Για τον, αντίκτυπο, τον αμυντικό αντίκτυπο του Brexit δεν είναι κάτι που συζητήθηκε. στην FAC. Οι συζητήσεις του Brexit λαμβάνουν χώρα εντός της ε, Task Force 50 του πλαισίου αυτού και εξ όσων γνωρίζω εκτός του πλαισίου αυτού δεν έχουν λάβει χώρα συζητήσεις. Για την άλλη σας ερώτηση δεν είναι τη αρμοδιότητός μου. Ε, ε, και προφανώς ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, έδρασε με βάση την δική του κρίση δεν είναι ούτε η αρμοδιότητά μου ούτε η θέση μου να σχολιάσω την επιστολή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θα έλεγα και κάτι άλλο αλλά σταματώ για το Αθήνα και το ICSP που αναφερθήκατε. Έχουμε δει τους περιορισμούς στην στήριξη που μπορούμε να παρέχουμε ε, στον εξοπλισμό ή και στην κατάρτιση στρατιωτικών ε, μονάδων μέσω του προϋπολογισμού του 41-2 επιβάλλει περιορισμούς. Υπάρχουν και ερμηνείες της νομικής αυτής διατάξεως που περιορίζουν τη δυνατότητα δράσεως εντός του προϋπολογισμού. Κοινή ερμηνεία, αν θέλετε, όλων είναι ότι πρέπει να εξετάζει κανείς ε, δημοσιονομικούς, ε, μάλλον χρηματοδοτικούς πόρους εκτός προϋπολογισμού Βεβαίως γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν που υφίστανται τεράστιες δημοσιονομικές πιέσεις και αυτό το βλέπουμε στις αποστολές κατάρτισης εκπαίδευσης ότι θα μπορούσαμε περισσότερο να βοηθήσουμε στα εξοπλιστικά, θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πρέπει να βρούμε επαρκείς ε, ε, χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Η πρόταση που προετοιμάζεται και είναι πρόταση απλώς και συζητείται ανοιχτά θα συνδύαζε σε μία facility τις δικές μας θεατρικές επιχειρήσεις υπό το CSDP, υπό το Αθήνα, με δράσεις που αυτή τη στιγμή ε, χρηματοδοτούνται από την Αφρικανική Facility για την Ειρήνη και άλλες δράσεις που δεν χρηματοδοτούνται, τμήματα του CPSD που δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε από τον προϋπολογισμό. Βέβαια όλα αυτά που σας λέω συζητούνται, δεν μπορώ να πω για πόσο καιρό θα συζητούνται και πόσο λεπτομερείς θα είναι οι προτάσεις και πότε αυτές θα υποβληθούν. Αλλά αυτό που λέτε δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα, αν θέλετε, ή την πρόθεση. Βεβαίω τα κράτη-μέλη τελικώ θα αποφασίσουν αν του ενδιαφέρει ή όχι να γίνει υπό την Αθήνα αν θα δημιουργεί μια άλλη facility θα ήταν κανονικά κάτι καινούριο. Αυτό που θα μας βοηθούσε να ξεπεράσουμε δηλαδή τους περιορισμούς που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον ε, Πρέσβη Επιτρέψτε μου να θέσω ένα συμπληρωματικό ερώτημα από την πλευρά μου, καθώς έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, τον οποίο θέλουμε να αξιοποιήσουμε για να συζητήσουμε περίπτωση μαζί σας. Ε, αναφερθήκατε στις σημαντικές αποφάσεις που ελήφθησαν σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την ε, παράταση των ε, project στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθωμένης συνεργασίας. Μήπως θα μπορούσατε να αναφέρετε τα πιο ενδιαφέροντα από αυτά. Από τη δική σας οπτική γωνία; Ναι, νομίζω πως αυτά τα project ε, σε αυτή τη φάση καθορίζονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια αυτή την περίοδο. Οπότε θα πρέπει να αναμείνουμε τον καθορισμό τους. Κάποια από αυτά έχουν πιο επιχειρησιακό χαρακτήρα ε, και προσπαθούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις ικανότητες μας σε επίπεδο επιμελητίας, σε εφοδιαστικής, σε επίπεδο ιατρικής περίθαλψης. Ε, στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο πλαίσιο της ανάπτυξης δυνάμεων. Άλλα project τώρα στοχεύουν σε μηχανισμούς ε, ε, ε, χωρίς εντολών και ελέγχου που στοχεύουν περισσότερο στον βιομηχανικό τομέα και υπάρχει και ένα project το οποίο για παράδειγμα αφορά στη δημιουργία ενός τεθωρακισμένου οχήματο. Δηλαδή υπάρχουν μία σειρά από διαφορετικά projects σε αυτό το τομέα και είναι σημαντικό τα υφιστάμενα project που ήδη τρέχουν να βοηθήσουν περισσότερο στην ομάδα, στην, στην εφαρμογή στην πράξη αυτή τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία. Ε, και από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουμε να εξετάζουμε και σε πιο ε, λεπτομερή βαθμό το τι ακριβώς θα χρειαστούμε στο επίπεδο αυτών των project καθώς ε, θα έχουν και άμεσα επιπτώσεις στο CPD, δηλαδή στο σχέδιο σε ό,τι αφορά τις ε, ικανότητες ανάπτυξης ε, δυναμιού. Άρα λοιπόν είναι καλό το ότι έχουμε ε, εδώ project και των δύο τύπων, δηλαδή project τα οποία μπορούν να έχουν επιχειρησιακή εφαρμογή άμεσα, ενώ κάποια άλλα θα είναι εκείνα που θα δώσουν τα αντίστοιχα ενάβσματα στη βιομηχανία για ανάπτυξη δηλαδή προς εκείνη την κατεύθυνση. Από τα 17 συνολικά project, 5 έως 6 είναι υποψήφια προς χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Πράγμα το οποίο αυτό καθεαυτό είναι θετικό. Αλλά όπως είπα βρισκόμαστε ακόμα στα πρώιμα στάδια αυτών των ε, project του σχεδιασμού τους και νομίζω πω ε, ε όσοι προτείνουν αυτά τα project θα τα ε, παρουσιάσουν με περισσότερες λεπτομέρειες και θα τα ορίσουν καλύτερα μέσα στις ερχόμενε εβδομάδε. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Ο κύριο Πασκού θέλει να θέσει κάποιο ερώτημα ακόμα. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, παρουσίαση και για αυτή την ε, πρωτοβουλία σας ε, να μας κρατάτε ενήμερους ως προς τις εξελίξεις. Το ερώτημά μου εμένα θα ήταν το εξής. Μας είπατε πως υπάρχει πλήρης ευελιξία σε ό,τι αφορά την ενεργοποίηση του άρθρου 42 παραγραφός 7. Νομίζω πως η Γαλλία το έκανε σε ό,τι αφορά το έρμπασε και σε σχέση πάντοτε με την ρήτρα αλληλεγγύης. Αυτή λοιπόν η ευελιξία του 42 7 θα διατηρηθεί. Α πούμε ότι αύριο θα υπάρξει μια άλλη χώρα η οποία θα θελήσει να ενεργοποιήσει τη διαδικασία του 42. Ε, θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα εντό εισαγωγικών το οποίο έθεσε η Γαλλία, το προηγούμενο δηλαδή αυτό της Γαλλίας ή όχι. Γιατί θα θυμόσαστε ότι το 2012 είχαμε συντάξει μια έκθεση ό,τι αφορά αυτές τις δύο ρήτρε, δηλαδή της αλληλεγγύης και της υποστήριξη, ε, και είχαμε αναφέρει ότι ενδεχομένως να συντηθεί ή στο μέλλον και πάλι η ενεργοποίηση αυτών των ρητρών. Ε, και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό το ενδεχόμενο, γιατί αποτελεί βέβαια προνόμιο των ε, κρατών μελών. Αυτό δηλαδή που θέλω να διασφαλίσω είναι ότι αν ένα κράτο μέλο ενεργοποιήσει την λόγω διαδικασία δεν θα δεσμεύεται από το προηγούμενο τη Γαλλία. Ναι, ευχαριστώ. Συμφωνώ πλήρω με τα όσα είπατε. Ναι, δεν θα υπάρξει τέτοιο προηγούμενο του πράγμα τη Γαλλία. Δηλαδή, αυτή είναι και μία από τι βασικέ αιρετέ αυτού του άρθρου. Δεν υπάρχει δηλαδή μία συγκεκριμένη διαδικασία, δεν υπάρχουν ε, κανόνες που προβλέπονται. Κάθε φορά η ενεργοποίηση εξαρτάται από το αίτημα του κράτους μέλους εκείνο το οποίο ενεργοποιεί το άρθρο και αξιώνει υποστήριξη. Και νομίζω πως και στη διατύπωση του άρθρου αναφέρεται αυτό με όλα τα δυνατά μέσα, with all possible means. Κατά συνέπεια, λοιπόν, το κράτος μέλος που ενεργοποιεί τη διαδικασία του άρθρου 42 έχει την ευελιξία να ζητήσει το είδος της αλληλεγγύης που εκείνο επιθυμεί, ανάλογα με τι ιδιαίτερε περιστάσει και ανάλογα ε, με αυτό που θα ζητήσει. Εάν ε, θέλαμε να θεσπίσουμε τόσο συγκεκριμένου κανόνες, ουσιαστικά θα δημιουργούσαμε μεγάλη σύγχυση. Θα ξεκινούσε μια τεράστια συζήτηση ανάμεσα στα διάφορα θεσμικά όργανα του Συμβουλίου, πράγμα στο οποίο βέβαια είμαστε συνηθισμένοι, αλλά τελικά δεν θα καταλήγαμε και σε ένα πιο χρήσιμο εργαλείο. Ένα από τα βασικά ρήματα αυτού του εργαλείου είναι ακριβώς η ευελιξία του, βέβαια, αλλά αυτή είναι η δική μου θέση ο κύριο ο κύριος Πασκ. Ναι, η Γαλλία είναι μια μεγάλη δύναμη, αυτό θέλω να πω, και όλοι θέλουν να την υποστηρίξουν. Αλλά αν πρόκειται για μια μικρότερη χώρα η οποία θα ήθελε να επαναλάβει αυτή τη διαδικασία, θα λάμβανε την ίδια αντίδραση. Ναι, όταν είχε ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, ανακοπήθηκε δηλαδή το άρθρο από τη Γαλλία, ήταν εντυπωσιακή η ανταπόκριση των πολυμοκρατών μελών. Ναι, εντάξει, εκεί πραγματικά υπήρξε αυτή η αλληλεγγύη, λέει ο κ. Πάσχου, γιατί ε, το αίτημα έγινε και αμέσω μετά τι δημοκρατικέ επιθέσει. Ναι, αυτή η ίδια αλληλεγγύη θα επιδειχθεί εάν ε, η διαδικασία δεν ενεργοποιηθεί από άλλο κράτο μέλο. Υπάρχει δηλαδή αυτό το δικαίωμα για όλα ε, τα κράτη-μέλη και δεν προβλέπονται συγκεκριμένε διαδικασίε. Οπότε δεν βλέπω το γιατί να υπάρξει διαφορετική διαδικασία στο μέλλον, αλλά βέβαια δεν μπορώ να είμαι σίγουρο γιατί μπορούν να υπάρξουν εκπλήξεις ε, στο μέλλον. Ναι, ε, εγώ θα ήθελα να επαναλάβω το αρχικό ερώτημά μου. Δεν νομίζετε πως θα πρέπει να προσαρμόσουμε το άρθρο 42 παράγραφος 7 ε, προκειμένου να ανταποκρίνεται στα νέα είδη απειλών, για παράδειγμα στις νέου είδους κυβερνοεπιθέσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως είναι διατυπωμένη 7η παράγραφος, αναφέρεται σε θύμα ένοπλης επίθεση, δηλαδή armed aggression. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν αναφέρεται στα νέα ίδια απειλών τα οποία αντιμετωπίζουμε σε ψηφιακό επίπεδο, σε κύβερνο επίπεδο και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν το ερώτημά μου είναι δεν θα πρέπει να προσαρμοστεί αυτό το άρθρο στις νέες απειλές, στους νέους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Κύριε Πρέσβη. Ναι. Όλοι μπορούμε να έχουμε τη δική μας άποψη σε σχέση με αυτό το ζήτημα μπορούμε να κάνουμε και μια επιμακρόν συζήτηση ως προς το αν αυτές οι επιθέσεις στο κυβερνοχώρο θεωρούνται τελικά ένοπλες επιθέσεις ή όχι. Κατά τη δική μου άποψη, ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα αυτού του άρθρου είναι η ευελιξία του και από εκεί και μετά υπάρχουν μια σειρά από διαφορετικοί μηχανισμοί για την επίδειξη αλληλεγγύης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η δική μα άποψη. Και γνωρίζετε βέβαια και ποιε είναι οι δυσκολίε, αν θέλει κανεί να τροποποιήσει τι συνθήκε. Έχουν ξεκινήσει ολόκληρε συζητήσει σε ό,τι αφορά το κυβερνοχώρο και συζητήσει επί τη αρχή, δηλαδή του κατά πόσο μια κυβερνοεπίθεση και πότε θα μπορεί να λογίζεται ως ένοπλη επίθεση ή όχι και νομίζω πως αυτή η οχι και νομιζω πω αυτη η συζητηση θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Και όπω είπα δεν μπορώ εγώ να αποφασίσω αν το άρθρο αυτό χρήζεται περαιτέρω τροποποίηση ή όχι. είναι περιορισμένη η διατύπωσή του, έχει λίγες λέξεις, οπότε δεν μπορώ να προσθέσω κάτι ακόμα. Ε, όλοι έχουμε διαφορετικές απόψεις και κάθε μία από αυτές είναι σεβαστή. Σας ευχαριστώ. Ε, Κύριε Πρεσβευτά, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων πριν την άρξη της συνεδριασής μας, Είπατε ότι θα θέλατε ίσως να σχολιάσετε κάποια θέματα που αφορούν τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ και είχαμε την παρουσίαση του προγράμματος που νομίζω ξεκίνησε η Λιθουανία και που παρουσίασε ένας διπλωμάτης Λιθουανός από τη μόνιμη αντιπροσωπεία τους. Και είχαμε ακριβώς τη συζήτηση για το σχέδιο της ΠΕΣΚΟ για την ομάδα ταχείας αντίδρασης στον κυβερνοχώρο. Και υπήρχαν κάποια ερωτηματικά ή παρατηρήσεις σε σχέση με τις δυνατότητες που υπάρχουν σε αυτό το επίπεδο για να ληφθεί υπόψη η συνεργασία ΝΑΤΟ-ΕΕ. Αλλά φαίνεται ότι σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή συνεργασίας μεταξύ των χώρων μελών, είναι δύσκολο να υπάρχει αυτή η σύνδεση με το ΝΑΤΟ. Υπάρχει κάποια δυσκολία από ό,τι φαίνεται. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα και συνεργασία στον κυβερνοχώρο νομίζω ότι είναι ένα από τα εξέχοντα σημεία συνεργασία και των δύο οργανισμών. Οπότε εμείς πώς θέλουμε να προχωρήσουμε εδώ τα πράγματα και ποια είναι τα επόμενα βήματα που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη εδώ. Όπω λέγατε και εσείς, ο κυβερνοχώρος όντω είναι ένα θέμα συνεργασίας και συζητήθηκε ένα από τα κυριότερα θέματα, α πούμε, είναι η κατανομή και στην προηγούμενη διαδικασία καταλήξαμε μια κοινή δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ και των δύο Προέδρων. Οπότε όντως αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό όπω είδαμε με τις ε, πρόσφατες κρίσεις και εκεί μπορούν να συνεργαστούν οι δύο οργανισμοί. Και είναι σημαντικός βέβαια και ο ρόλος των ομάδων που ασχολούνται με αυτό. Σημαντικό το θέμα επίση τη κατανομή πληροφοριών μεταξύ των οργανισμών και αυτό σχετίζεται και με εσά. Τώρα, κατά πόσο το προσωπικό μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω, αυτό είναι άλλο ζήτημα, να το έχουμε αυτό κατά νου, γιατί πραγματικά αφορά διάφορες μορφές συνεργασίες. και δεν χρειάζεται, μάλλον δεν σχετίζεται και τόσο με την πραγματική καθημερινή συνεργασία μεταξύ των εργασίων. αλλά αυτό είναι, ξαναλέω, πρόβλημα άλλης φύσης και επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο συντονίζουμε τις απαντήσεις μας και συνεργαζόμαστε. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι. Δεν βλέπω άλλε παρατηρήσει. Ε, Σα καλώ να χειροκροτήσουμε θερμά τον κύριο Πρέσβη και να πω ότι εμείς βασιζόμαστε στην παρουσία σας και στην ενημέρωσή σας μετά από τα Συμβούλια Ασφάλειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, χαρά μου, χαρά μου που βρίσκομαι εδώ, λέει ο κ. Πεσβευτή. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, λέει πρόεδρο, στις 5 θα έρθουν οι εμπειρογνώμονέ μα οπότε θα πρέπει να διακόψουμε μέχρι τις 5 το απόγευμα και μετά θα έχουμε τη συζήτηση που θα αφορά την ασφάλεια στο Αφγανιστάν σε συνεργασία με την αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν. Συνάδελφοι, παρακαλώ να καθίσετε γιατί έχουμε φτάσει στο τελευταίο σημείο για σήμερα έχουμε άλλη μισή μέρα αύριο το θέμα λοιπόν για τώρα είναι η κατάσταση ασφαλείας στο Αφγανιστάν ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Πέτρα Όστρεβιτς που είναι επικεφαλής της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν Επίσης να σας παρουσιάσω τα υπόλοιπα μέλη του πάνελ ο κύριος Δίτμα Κρίσλα επικεφαλής της μονάδας της ΙΕΔ που ασχολείται με Αφγανιστάν και Πακιστάν. Στα αριστερά μου ο κύριος Μάρτιν Τιπάολο που είναι υπεύθυνος για θέματα που αφορούν στο Αφγανιστάν και το Ιράκ ή στο ΝΑΤΟ επικεφαλής των επιχειρήσεων πολιτικής έκανε ένα σφάλμα η πρόεδρος και το διόρθωσε Αφγανιστάν και Ιράκ λοιπόν επίσης έχουμε τον πρέσβη Μπάτου Κουτέλια πρώην πρέσβη της Γεωργίας στι Ηνωμένε Πολιτείε και μέλος στο Ερευνητικό Ινστιτούτο McCain στο Πανεπιστήμιο του Arizona State και βεβαίως η κυρία Ντογοτέ Βοντάμ του Καθολικού Πανεπιστημίου της Λουβά όπου συμμετέχει και αυτή σε, ως επίκουρος καθηγήτρια στη μελέτη κρίσεων και διεθνών αντιπαραθέσεων του Πανεπιστημίου του Λουβά. Να θυμίσω τώρα στον συνάδελφο κύριο Στρεβίτσιος ότι έχουμε τέσσερις ομιλητές και επομένως παρακαλώ να είστε όσο πιο σύντομα γίνεται. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είχαμε πολλές συναντήσεις ε, σήμερα, δεν πρόκειται να σας κουράσω με μακροσκελή εισαγωγικά σχόλια. Ευχαριστώ πάντως συνάδελφοι. Ευχαριστώ τους προσκεκλημένους εκ των προτέρων για την συζήτηση που θα έχουμε για το σημερινό θέμα που δεν είναι καθόλου βαρετό. Η κατάσταση της ασφαλείας στο Αφγανιστάν και ευχαριστώ και όλα τα μέλη της Επιτροπής Τώρα να πω ότι η πρώτη εξέλιξη είναι μια αρνητική εξέλιξη στην ασφάλεια που βασίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία. Να αναφέρω απλώς ότι το 2017 είχαμε 57 επιθέσεις αυτοκτονίας με 605 θύματα, νεκρούς δηλαδή, και ε, περί τους 1.900 τραυματίες. Τον Ιανουάριο μόνο φέτος είχα μια σειρά επιθέσεων 20 Ιανουαρίου με 22 νεκρούς 24 Ιανουαρίου 6 νεκρούς 27 Ιανουαρίου εκρήξεις με τουλάχιστον 100 νεκρούς 29 Ιανουαρίου 11 στρατιώτες από επίθεση της ISIS λέει ο μελτής Κάποιοι λοιπόν γνώστες της κατάστασης εκεί λένε ότι οι Ταλιμπάν απειλούν περί το 70% της επικράτειας του εδάφους. Κάποιες ομάδες των Ταλιμπάν διαβιβάζουν το μήνυμα ότι θέλουν να τελειώσουν τον πόλεμο, ότι θέλουν να εκκινήσουν διαπραγματεύσεις. Η κυβέρνηση του Αφγανιστάν έχει κάνει κάποιες παραχωρήσεις, κάποιες υποχωρήσεις οι νέες προσφορές ειρηνευτικών συζητήσεων συνοδεύονται από ενισχυμένη αμερικανική αποστήριξη ώστε να μην έχουν περαιτέρω ανάκτηση στα Ταλιμπάν που θα μπορούσε να είναι ένας από τους λόγους που λένε ότι θέλουν ειρηνευτικές συζητήσεις ώστε να πιστούν ότι δεν μπορούν να κερδίσουν τον πόλεμο. κύριος Πριζιντάνη λέει ότι θέλει να απευθυνθεί στο σύνολο των Ταλιμπάν, αλλά η ηγεσία τους είναι τόσο κατακαιρματισμένη που είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς συνομιλητές όπου θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν μια βάση του πυρός. Και στο πλαίσιο αυτό, το δύσκολο αυτό, περίπλοκο πλαίσιο που ισχύει στο πεδίο, περιμένουμε ενδιαφέρον τη σημερινή συζήτηση για να έχουμε περισσότερες πληροφορίες, επικαιροποιημένη ενημέρωση για την κατάσταση που ισχύει σήμερα στο έδαφος. Λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστέρηση λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον κύριο Κρίσλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες ε, απόψεις αναλύσεις της ΙΕΔ. Πράγματι έχει δυσχεράνει σημαντικά η κατάσταση της ασφάλειας ε, στο Αφγανιστάν. Οι επιθέσεις και στην Καμπούλ και στην Τζαλαλαμπάν του Ιανουαρίου απλώς το καταδεικνύουν αυτό. Σύμφωνα με την τελευταία μεγέθη του Ιανουαρίου 16 είναι αυτά. Ο έλεγχος της ε, αφγανικής κυβέρνησης επί των τμήματων του εδάφους είναι ο πιο χαμηλός. Οι ανταρτικές ομάδες έχουν τον υψηλότερο έλεγχο από το Δεκέμβριο του 2015. Η πλειοψηφία των ε, επαρχιών υπό τον έλεγχο των εξεγερθέντων έχει διπλασιαστεί. Και οι επαρχίες που στις οποίες αντιμάχονται οι δυνάμεις έχουν αυξηθεί κατά 50%. Τα τμήματα εκείνα λοιπόν της χώρας που ελέγχει η αυγανική κυβέρνηση έχουν μειωθεί κατά άνω του 20%. Όλα αυτά μας δείχνουν με συντομία την δυσχεράνουσα αυτή κατάσταση. Τώρα, στην τελευταία συνάντηση της λεγόμενης Kabul ε, Process, στο τέλος περασμένου μήνα, η Αφγανική κυβέρνηση υπέβαλε μία άνευ προηγουμένου πρόταση ειρήνης, προσφορά ειρήνης προς τους Ταλιμπάν. Ο, ο πρόεδρος Γκάνι περιέγραψε την ε, πρόταση ως μεγαλύτερη ελπίδα που υπήρξε τα τελευταία 18 χρόνια. Με εισαγωγικά αυτό. Μεταξύ της πρότασης πάυση του πυρός και απελευθέρωση εχμαλώτων, νέες εκλογές που θα συμπεριλαμβάνουν τις ένοπλες ομάδες και πρόταση ειρήνης προς τους Ταλιμπάν. και εμείς ελπίζουμε ειλικρινά ότι αυτή η πρόταση θα γίνει αποδεκτή από, το Ταλιμπάν, από τους Ταλιμπάν ώστε να οδηγηθούμε σε μια γνήσια ειρηνευτική διαδικασία αλλά δεν υπάρχει καμία σαφήνεια, καμία ασφάλεια ως προς το πώς θα ανταποκριθούν, πώς θα αντιδράσουν οι Ταλιμπάν έναντι αυτού. Δεν έχουμε δει κανένα είδους επίσημη απάντηση. Είναι δεν είναι ιδιαίτερα πιθανό ότι θα μειωθούν τα φαινόμενα βίας και πάρα πολλές ένοπλες ομάδες θα μπορούσαν να παρέμβουν σε οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία και οι λεγόμενοι ομάδες ε, οι πιο σκληροπυρηνικές όπως και τα στοιχεία της Daesh ISIS που έχουν διεισδύσει λέει ο μιλητής στη χώρα άλλο είναι ερωτηματικό είναι οι μελλοντικέ ε, πράξεις του Πρόεδρου Γκάνη. Του χρόνου θα υπάρξουν εκλογές και θα είναι υποψήφιος μάλλον, αλλά παράλληλα θα έχει να αντιμετωπίζει έντονη πίεση, απειλές δηλαδή για την ασφάλεια. Δεν γνωρίζουμε πώς θα μπορέσει πώς τελικώς θα αντιδράσει απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα και απέναντι στην κοινή γνώμη. Και υπάρχει και μια σειρά διεθνών δυνάμεων και φορέων που θα πρέπει να τοποθετηθούν. Ευθυγραμμιζόμενοι ή όχι προς την πρόταση ειρήνευσης του Γκάνη. Μιλώ για το Πακιστάν, αλλά μιλώ και για την Ρωσία και το Ιράν. Πρέπει πάντως να διατηρηθεί αυτή η όθηση προς τα εμπρός. Και μια σημαντική συνάντηση στην Τασκένδη στο Ουσμπεκιστάν την ερχόμενη εβδομάδα 26-27 Μαρτίου θα λάβει χώρα και θα είναι μια σημαντική ευκαιρία να ε, επαναληφθεί, να επανυπογραμμιστεί η διεθνή στήριξη προς την πρόταση του Πρόεδρου Γκάνη. Προσπαθώντας να αποστείλουμε σημαντικό μήνυμα από τη διεθνή κοινότητα αλλά και προς τους Ταλιμπάν ότι πρέπει να ανταποκριθούν στην ειρηνευτική προσφορά του Πρόεδρου Γκάνη και ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία αυτή να εισέλθουν σε μια ειρηνευτική διαδικασία. Για τα επόμενα βήματα λοιπόν να πω ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι η διεθνή κοινότητα θα, θα εργαστεί, θα συνεργαστεί πιο συλλογικά, ότι θα συντονιστεί καλύτερα και ότι θα συμφωνήσει προς κοινά μηνύματα προς τους Ταλιμπάν, αλλά και προς το Πακιστάν. Ότι η διεθνή κοινότητα θα μειώσει τον αριθμό των οντοτήτων των φορέων που μιλούν με τους Ταλιμπάν, διότι αυτό δημιουργεί σύγχυση και σε κάποιο βαθμό τους ενισχύει. Και πάρα πολλοί φορείς της διεθνούς κοινότητας μιλούν του Ταλιμπάν. Θα ήταν σημαντικό να συνεδευτεί επίσης η ειρηνευτική διαδικασία με πολιτικά μέτρα, χωρίς πίεση προς το Ταλιμπάν, αλλά με συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να είναι επιπαραδείγματοι. Η σύσταση ούτως αποκαλούμενων ασφαλών ζωνών, safe zones για να συνεννοούμεθα, οι οποίες θα παρουσιάζονταν ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης και προς την ειρήνη, δηλαδή στην ουσία περιοχές τοπικής πάυσεως του πυρός προς την ε, προστασία και ασφάλεια των κατοίκων των περιοχών αυτών. Και η διεθνώς κοινότητα θα πρέπει να είναι έτοιμη να παράσχει υποστήριξη για τέτοια μέτρα. Θα ήταν επίσης σημαντικό να δει κανείς τι θα έπρεπε να έλθει μετά, επόμενο σε μια ειρηνευτική διαδικασία και θα μπορούσαμε να εμπνευστούμε από περιπτώσεις όπως η Κολομβία, η Συρία σε κάποιο βαθμό λέει ο μίλητης, αλλά και Βαλκάνια όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε θεμελιώδου σημασία ώστε να υπάρξει μια συμφωνία με την, ομάδα Hesby Islami Έχουμε, υποστηρίζουμε λοιπόν αυτήν την διαυγανική ειρηνευτική πρόταση που έχει τεθεί και επίσης θα ήταν σημαντικό να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σε έργα περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης και θα αναφερόμουν στην, ε, στο έργο του αγωγού του ΤΑΠΗ ή Κάζα ε, είναι έργα που είναι σημαντικά, τα αναφέρω ως παραδείγματα γιατί είναι σημαντικά για το πώς οι περιφερειακοί φορείς μπορούν να εμπλακούν, να συμμετάσχουν σε μία διαδικασία που οδηγεί προς την ειρήνευση γιατί ενισχύει την περιφερειακή ε, ολοκλήρωση και αποτρέπει τη συνέχιση των εχθροπαραξιών. Ευχαριστούμε τον κύριο Κρίσλα, ο κύριος Ντιπάολο τώρα, του ΝΑΤΟ. Thanks very much. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο Ευρωκοινοβούλιο. Είμαι από τους λίγους Αμερικανούς που ξέρουν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο και από τους ακόμα λιγότερους που έχουν πάει. Χαίρομαι πολύ που μιλάω στο τέλος μιας μακράς ημέρας σε μια ομάδα ατόμων που ενδιαφέρονται για το θέμα και αν σας ενδιαφέρουν αυτά που κάνουμε εκεί, υπέρ ή κατά, να έχει σημασία, είστε κατάλληλοι. Οπότε σας ευχαριστώ για την πρόσκληση θα βάλω τα δυνατά μου να με θυμάστε και να πω κάτι ουσιώδος και επίσης να τηρήσω το χρόνο των πολλών και θαυμάσιων ε, δημένων που έχετε δώσει νέους και το οποίο είναι νέο για μένα. Να πω καταρχάς ότι ήμουν πιλότος ελικοπτέρων και αυτό δεν το κάνεις με αισιοδοξία πρέπει συνέχεια να ρωτάς τον εαυτό σου τι χειρότερο θα μπορούσε να μου συμβεί τώρα. Αυτό πρέπει να το έχει παντά κατά νου. Και το ίδιο εφάρμοσα και στη δουλειά μου στο Αφγανιστάν. Πράγματι νομίζω ότι η αισιοδοξία είναι κατά πάσα πιθανότητα η, υπερφιλο, η συγγνώμη, είναι μία από τις ενδεχόμενες προσεγγίσεις του Αφγανιστάν αλλά το χειρότερο είναι ο κινησμός και είναι εύκολο να το κάνεις αυτό γιατί με κάποιες ασχημές ειδήσει το δικαιολογείς αλλά δεν σε οδηγεί σε κάποια επιτυχία. Η επιτυχία είναι το να σταθεί το Αφγανιστάν στα πόδια του και να υπάρχει ασφάλεια στην περιοχή. Δεν θα σα δώσω λοιπόν αισιόδοξη κοινική σκοπιά των πραγμάτων, αλλά θα ήθελα απλά και μόνο να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας. Η ασφάλεια είναι ξεκάθαρα χειρότερη, σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι πριν χρόνια. Συμφωνούμε γι' αυτό. Υπάρχουν πιο απτοί φραγμοί, μεγαλύτεροι, εντονότεροι, υψηλότεροι. Υπάρχει ένταση στις πόλεις δεν φαίνεται άμεσα γιατί υπάρχουν φραγμοί, αλλά έχει επιδεινωθεί η ασφάλεια. Έχουμε τον έλεγχο της κυβέρνησης που δεν είναι αυτός που πρέπει. Όταν είχαμε κάνει τη μετάβαση στο ΝΑΤΟ στις επιχειρήσεις μας ε, σε αποστολή υποστήριξης είχαμε αύξηση των θυμάτων μεταξύ του, των πολιτών και ο κ. Νίκολσον είχε πει ότι πραγματικά έχει βαλτώσει εδώ πέρα η κατάσταση και αυτά είναι τα δεδομένα λοιπόν. Και οι λογικοί άνθρωποι, άνθρωποι υπεύθυνοι όπως εσείς, άκουσαν για επιτυχίες, ε, ενδεχόμενες επιτυχίες επιτυχημένων δικητών στο Αφγανιστάν. Όταν δηλαδή οι Αφγανοί περιμέναμε να προχωρήσουν Οπότε οι λογικοί άνθρωποι τώρα αναρωτιούνται γιατί έχουμε βαλτώσει, γιατί εμείς συνεχίζουμε την, και εντείνουμε την παρουσία μας στην περιοχή και θα απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα. Τι έχει αλλάξει λοιπόν σε σχέση με τα προηγούμενα 16 χρόνια. Καταρχάς η νοοτροπία μας είναι διαφορετική. Μέχρι το 2014 προσπαθήσαμε να βάλουμε ε, μπροστά τους Αφγανούς. Αλλά τα προβλήματα παρέμειναν επειδή τα διακυβόμενα, διακυβευόμενα ήταν υψηλά. Και αν οι Αφγανοί απέτυχαν, εμεί ήμασταν εκεί για να τους βοηθήσουμε και να λύσουμε τα προβλήματα. Αυτό δεν το κάνουμε πια. Οι Αφγανοί είναι μόνοι του. Υπάρχει αρρωγή, εκπαίδευση κτλ. από το ΝΑΤΟ, αλλά δεν προσπαθούμε άμεσα ήδη να λύσουμε τα προβλήματα και είναι σημαντική η πρόοδο. Δεύτερον, η δικιά του νοοτροπία έχει αλλάξει. Όταν εμεί πήγαμε από την ISAF σε επιχείρηση υποστήριξη, υποστηρικτική, τότε αυτό αποτέλεσε ένα σημείο καμπή για του Αφγανού. Θα μπορούσε κανεί να πει, αν είμαστε ειλικρινεί εδώ, θα μπορούσαμε να πούμε και να παραδεχτούμε ότι το ΝΑΤΟ και η ΙΠΑ ίσω έκαναν πολλά και πολύ γρήγορα και αυτό θα μπορούσαν να το χαρακτηρίσουν κάποιοι ως μια κατάσταση ασφάλειας που χειροτερεύει. Χειροτέρεψε και έφτασε σε ένα επίπεδο σταθερότητας. Δεν χειροτέρεψε πολύ. Και τουλάχιστον βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου αναγνωρίζουμε τι συμβαίνει με την ασφάλεια στο Αφγανιστάν, όπου το ΝΑΤΟ και η ΕΠΑ δεν ασχολούνται με την ασφάλεια σε κάθε σημείο. Οπότε η δική μας νοοτροπία έχει αλλάξει και μετά από αυτή τη μεταβατική περίοδο, όπου είχαμε απώλειες, των κεκτημένων μας, βλέπουμε να ενισχύεται η αυτοπεποίθηση των Αυγανών και αυτό είναι νομίζω το μυστικό συστατικό που θα οδηγήσει την επιτυχία στο Αυγανιστάν. Και είναι δυσάρεστο, αλλά θα το πω ξεκάθαρα, η αποτελεσματικότητα και η εμπιστοσύνη, η αυτοπεποίθηση των Αυγανών μεταφράζεται στο κατά πόσο θανάσιμη είναι η δυνατότητα παρέμβασή του στα πεδία μάχη. Και αυτό είναι σημαντικό μετά από τόσα χρόνια συγκρίσεων. Είναι λοιπόν σημαντική η αυτοπεποίθηση των Αυγανών απαραίτητο συστατικό όταν ο Παραδός Κάνι έκανε μια θαραλέα ανεφόρον προσφορά για ερευνητικές διαδικασίε με τους Ταλιμπάν. Αν είχε αυτοπεποίθηση δεν θα το έκανε. Και τέλος, να σας πω ότι υπάρχει συνένεση στο Αφγανιστάν μεταξύ όλων των μπλεκομένων η Πανάτου, διεθνής κοινότητα, Αυγανών, ακόμα και τα Ταλιμπάν, ότι η στρατιωτική νίκη είναι αδύνατη. Δηλαδή βρισκόμαστε σε μια στασιμότητα αμοιβαία εξόντωση. Και εδώ δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ χρήσιμα να τα έχουμε κατά νου. Αν λοιπόν βελτιωθούν οι προϋποθέσεις επιτυχίας, αν είμαστε πιο ειλικρινείς για το πού βρισκόμαστε και αν έχουμε στερεότερη βάση, τότε ας δούμε ποια θα ήταν η πιθανή επιτυχία. Καταρχάς, το να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να υπάρχει αποδοχή κάποιων δεδομένων. Αν δείτε, ας πούμε, τον χάρτη του Αφγανιστάν, τον οικονομικό, αν δείτε, ας πούμε, ε, την εξέλιξη του ΑΕΠ, θα δείτε ε, ότι σχετίζεται με την, εξέλιξη, με την παρουσία του ΝΑΤΟ. Οπότε η κατάσταση αυτά είναι τεχνητή και παραμένει τεχνική σήμερα. Από το 9 μέχρι το 12, 2009 μέχρι το είχαμε αύξηση του ΑΕΠ κατά 12% και τώρα είμαστε στο 3%. Οπότε ρωτάω τι είναι πιο ρεαλιστικό και βιώσιμο και ότι είναι και πιο ειλικρινές ως αποδοχή. Ο Εθνικός Αμερικανικός ε, Στρατός προχωράει παντού. Όλα τα έξι σώματα στρατού βρίσκονται ε, σε προχωρημένη φάση. Έχουν προχωρήσει δηλαδή στις επιχειρήσεις τους. Αυτό είναι σημαντικό. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν περίπλοκες κοινέ επιχειρήσεις που εμπλέκουν ειδικέ δυνάμει, τακτικέ δυνάμει στρατού και άλλε δυνάμει. Όλε μαζί. Και αυτό είναι πολύ περίπλοκο γιατί λένε πολλοί στρατιωτικοί ότι η το έχουν καταφέρει ακόμα καλά και σχεδιάζουν αυτέ τι επιχειρήσει οι Αυγανοί για την... να τι εκτελέσουν μόνοι του. Και αυτό δεν συνέβαινε παλαιότερα. Απόλυε στον άμαχο πληθυσμό. Ευαίσθητο θέμα αυτό και αποτελεί πηγή μεγάλης απογοήτευσης για το γεγονό ότι υπάρχουν, αλλά για πρώτη φορά από το 2012, όπως θα γνωρίζετε, οι απώλειες αμάχων στις συγκρούσεις έχουν υποχωρήσει. Στις 22 από τις 34 επαρχίες έχουν υποχωρήσει αυτές οι απώλειες. Γιατί μειώθηκαν επειδή καταρχάς η επαγγελματικότητα των Αυγανών και η ηγεσία η στρατιωτική μείωσε, κατάφερε να μειώσει τις απώλειες της συγκρούς κατά 37%. Αυτό όμω σημαίνει ότι οι Αφγανοί ηγέτε ε, ρηψοκινδυνεύουν και ότι επίσης ηγούνται των επιχειρήσεων αυτών με πιο ευφυή τρόπο ώστε να μειωθούν σημαντικά οι απώλειες των αμάχων. Είχαμε μια αύξηση 24% στις απώλειες των αεροπορικών δυναμίων όσον αφορά το σύνολο των ατόμων που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις, αλλά όσον αφορά τις συγκρούσεις από έτος σε έτος, ε, νομίζω φέτος είμαστε στα ίδια επίπεδα του περασμένου έτους, δηλαδή 68 και 69 αντίστοιχα. Αυτά παραμένουν σταθερά. Πρέπει όμως να έχουμε κατά νου ότι έχουν διπλασιάσει τις ευρωπαϊκέ του επιχειρήσεις. Οπότε έχουμε στην ουσία μείωση των απολύων των αμάχων μετά από αεροπορικέ επιχειρήσεις. Με την ε, βοήθεια βεβαίω του ΝΑΤΟ και πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα στους Αφγανού γι' αυτό. Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Να πω όμως ότι είχαμε και πρόσφατη νομοθεσία στο Αφγανιστάν με την αποστράτευση υψηλών ε, αξιωματικών του στρατού και αυτό είναι σημαντικό για, τον, για τους εξής λόγους. Καταρχάς, αυτοί που απομακρύνθηκαν ήταν αυτοί που επιβίωσαν από την σοβιετική εποχή. Έχουν λοιπόν σοβιετικού τύπου νοοτροπία που δεν προωθεί βέβαια την καινοτομία, προωθεί την ε, κεντρική διοίκηση, κεντρικό στυλ διοίκησης και αυτοί αποχωρούν. Έχω όμως και τη γενιά αυτή το να... που έχουν επιβιώσει μπορεί να σου μιλήσει στα αγγλικά αλλά και στα ρωσικά. Και είναι μια γενιά που αποδέχεται και την αποτυχία, όχι μόνο την επιτυχία. Δεν επιζητά μόνο την επιτυχία. Αυτοί αντικαταστάθηκαν λοιπόν από την επόμενη γενιά επαγγελματιών στρατιωτικών που είναι διατεθειμένοι να λάβουν τα ενία. Αυτό τι σημαίνει, όλα αυτά τι σημαίνουν. Σημαίνει ότι μετά από 16 χρόνια συγκρούσεων θα πρέπει να αναπτυχθούμε ότι έχουμε πετύχει. Α κάνουμε λοιπόν μια καταγραφή. Καταρχά, έχουν αναλάβει οι ίδιοι Αυγανοί, όπω είπα. Δεύτερον, πριν το 2001 είχαμε 900.000 αγόρια στα σχολεία και μηδέν κορίτσια. Τώρα έχουμε 9 εκατομμύρια παιδιά, πολλά κορίτσια. Πρόσβαση στην ε, περίθαλψη. Τώρα είμαστε στο 57% του πληθυσμού. Πολύ υψηλότερα από το 2002. Ενδιαφέρουσα στα στρατι... Ε, στατιστική επίσης το ότι η γονιμότητα των ανηλίκων κοριτσιών, των εφήβων κοριτσιών έχει μειωθεί στο ίμιση. Οπότε αυτά τα κορίτσια δεν χρειάζεται να μεγαλώνουν οικογένεια και να έχουν παιδιά, μπορούν να πάνε στο σχολείο. Επίση, ανθούν και τα ανεξάρτητα αυγανικά ΜΜΕ, να δεν δώσω και άλλου αριθμού, είναι πολύ σημαντικοί πάντω. Πάντω και τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει ε, να τα επενέσουμε για τη συμμετοχή τους και για, την, για τα επιτέματα αυτά τα τελευταία 16 χρόνια. επιτεύγματα που, που επιτεύχθησαν στα πλαίσια αυτής της αφγανικής ηγεσία στα θέματα ασφαλείας. Θα σας πω και δύο τελευταία λόγια και θα σταματήσω. Έχουμε αυτή την προσφορά για ειρήνη και θα συνεχίσουμε όμως να εργαζόμαστε στον τομέα της ασφάλειας ώστε να βοηθήσουμε τους Αφγανούς να έχουν αυτοπεποίθηση και να συμβάλλουν στην ειρήνη. Το 18 θα είναι δύσκολο έτος για τους Ταλιμπάν γιατί βρίσκονται υποπίεση σε όλη τη χώρα συνεχόμενη και θα παραμείνει συνεχής η πίεση προς αυτούς. Όσο πάμε προς το 19 το σταδικό μας δυναμικό, είπα, ΝΑΤΟ, τον ίδιο των Αφγανών οι Αφγανοί μάλιστα έχουν διπλασιάσει τον αριθμό των ειδικών δυνάμεων και έχουν τετραπλασιάσει μάλιστα ε, και τον αριθμό των αεροπορικών δυνάμεων. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι πάμε στο 19, 19 που θα είναι η πρώτη χρονιά που όλα αυτά τα εργαλεία θα εφαρμοστούν από κοινού κατά του κοινού εχθρού στο Αφγανιστάν. Το 19 λοιπόν θα είναι χειρότερο για τους Ταλιμπάν. Αν θα ήσασταν λοιπόν ηγέτης των Ταλιμπάν τότε έχει έρθει η ώρα να ρωτηθείτε αν πρέπει να συζητήσετε για ειρήνη και το 18 βεβαίω προσπαθούν να δουν κατά πόσο το 19 θα είναι χειρότερο αυτή. Οπότε εγώ προσβλέπω σε σημαντικές αλλαγέ όσον αφορά την σκοπιά των Ταλιμπάν μέχρι τα μέσα του 19 που ενδεχομένω θα αρχίσουν να, να παραδίδονται και να βλέπουν ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, άλλη διέξοδο για αυτού. Από τους συμμάχους που απαρτίζουν το ΝΑΤΟ βλέπουμε ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τις προσπαθίες μας στο πολιτικό σκέλος, όχι μόνο στο στρατιωτικό και ε, θα πρέπει να διευρύνουμε τις ε, δεσμεύσεις μας για επενδύσεις ε, πέραν των, του ορίζοντα χρονικού όριστου που έχουμε προκαθορίσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Μπάτου Κουτέλια. πρώην πρεσβευτή τη Γεωργίας στη ΣΥΠΑ και τώρα εμπειρογνώμονα στο Ινστιτούτο Μακέιν για την ειδική ηγεσία στο, στο Πανεπιστήμιο Πολιτεία Αριζόνα. Σα ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα εδώ και έχω την ε, δυνατότητα να συζητήσω μαζί σα ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα τη ε, Παγκόσμια ασφάλειας, δηλαδή αυτό το Αφγανιστάν. Και χαίρομαι επίση ε, που βλέπω μια κοινή συζήτηση από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το ζήτημα. Πραγματικά αυτό θα αποτελέσει το κλειδί για την ε, επιτυχία εκεί. Η αποστολή στο Αφγανιστάν είναι εξαιρετικά σημαντική για την ε, γεωργία, όχι μόνο γιατί είμαστε οι πιο σημαντικοί χορηγή σε ό,τι αφορά αυτή την επιστολή σε επίπεδο κατά κεφαλαία, αλλά επειδή είναι και τόσο σημαντική η κατάσταση του Αφγανιστάν για την ευρύτερη περιοχή. Ε, δύο ζητήματα θα θίξω καταρχήν την γενική κατάσταση σε αυτή την περιοχή και το πώς το Αφγανιστάν επηρεάζει ακριβώς την γενικότερη κατάσταση στην περιοχή και από εκεί και μετά θα αναφερθώ σε κάποιες πρακτικές επιπτώσεις, για κάποια πρακτικά εργαλεία τα οποία θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε ούτως ώστε οι διαδικασίες να κατευθυνθούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Όπω ήδη αναφέρθηκε από του προηγούμενου ομιλητέ, ε, το ζήτημα του Αφγανιστάν είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Έχουμε δηλαδή τη διάσταση τη ε, ασφαλεία, ε, τη Ανάπτυξη ε, και άλλων, αλλά τελικά σε τελική ανάλυση χρειάζεται μια συντονισμένη δράση από όλους τους κρατικούς εφορείς του Αφγανιστάν. Αλλά βέβαια το ζήτημα δεν είναι απλά και μόνο ζήτημα τεχνικής εκτέλεσης των διαφόρων απαιτούμενων μέτρων, αλλά είναι και ένα ζήτημα πολιτικής βούλησης. Τι θέλει να κάνει το Αφγανιστάν, ποιο ρόλο θέλει να παίξει στο μέλλον. Από ιστορικής άποψης, αποτελεί ένα δόγμα Τρούμαν αν θέλετε σε αυτή την περιοχή ότι δηλαδή υπάρχει ε, ένα στρατιωτικό μια στρατιωτική διάσταση και μια οικονομική διάσταση, όπως για παράδειγμα το σχέδιο Μάρσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν υπάρχουν αυτές οι δύο διαστάσεις και το τμήμα που λείπει εδώ είναι ακριβώς ένα πολιτικό όραμα, αυτή η διάσταση του πολιτικού οράματος για το Αφγανιστάν και νομίζω πως ε, και εμείς από την πλευρά μας διαπιστώνουμε πως υπάρχει αυτό το κενό, ότι δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η πολιτική ηγεσία. Άρα λοιπόν όταν δεν υπάρχει πολιτικό όραμα και ηγεσία τότε ε, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες έρχονται και πληρώνουν αυτό το ε, κενό. Πράγμα το οποίο βέβαια οδηγεί σε εκνομισμό. Ε, Παρ' όλα αυτά εγώ ε, είμαι και εγώ αισιόδοξο από την πλευρά μου, αξιολογώ τη σημερινή κατάσταση ως καλύτερη, καλύτερη Και ε, εντάξει μπορεί κανείς να έχει μια πιο αισιόδοξη, μια απεσιόδοξη ε, άποψη για τα πράγματα, αλλά ε, εξετάζοντας δυναμικά την κατάσταση διαπιστώνει κανείς πράγματι ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Και αυτό ε, αν το δούμε πιο μακροσκοπικά δηλαδή. Ε, τα όσα συμβαίνουν στο Αφγανιστάν θα πρέπει να ενταχθούν στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής και πολιτικής τη ε, Δύσης απέναντι στις χώρες της περιοχής όπως η ε, Ρωσία, η Κίνα, το Πακιστάν και η Βόρειος Κορέα. Άρα λοιπόν η πολιτική που ασκούμε στο Αφγανιστάν θα πρέπει να σχετίζεται άμεσα και με τη Ρωσία γιατί η Ρωσία θέλει να δημιουργήσει όσο μεγαλύτερη ζημιά και βλάβη γίνεται στην Δύση στο πλαίσιο του, του, του ντόγματος ε, του Πούτιν ε, κατά δηλαδή του δυτικού ελεύθερου κόσμου. Από εκεί και μετά υπάρχει ένα ακόμα τμήμα και αυτό είναι οι διάφορες ε, διαδικασίες συστομάτωσης αλλά και ε, κατακαιρματισμού σε διάφορα επίπεδα οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό. Ε, για παράδειγμα, ακούμε σε ό,τι αφορά αυτό το, την σύλληψη της μία σε ένας δρόμος, one belt, ε, one road που προωθεί ως όραμα η Κίνα στο οικονομικό επίπεδο. Το ΝΑΤΟ, οι δηλαδή σύμμαχοι Ευρώπης ε, και Αμερικής ε, είχαν ένα κοινό όραμα σε ό,τι αφορά το στατιστικό επίπεδο σε σχέση με την παράβαση στο Αφγανιστάν, αυτό το επωνομαζόμενο Northern Distribution Network ε, και το διαχωρισμό δηλαδή της χώρας σε ε, βορρά ε, και σε ό,τι αφορά την οργάνωση των επιχειρήσεων. Υπήρχε δυνατότητα να καταστεί επιχειρησιακή, επιχειρησιακό αυτό το, το δίκτυο με πρόσκληση δηλαδή και εταίρων από τη Δύση έτσι ώστε να υπάρξει μια σχέση η οποία θα απέφερε ωφέλη για όλες τις πλευρές προκειμένου δηλαδή να εκινηθεί και η οικονομία στο Αφγανιστάν με αυτόν τον τρόπο. Ε, υπάρχουν κάποια στοιχεία που στέφτηκαν με επιτυχία, αλλά θα χρειαστεί αυξημένη παρουσία από τη Δύση, από τις χώρες εταίρους, ε, στο πλαίσιο δηλαδή και του δρόμου του μεταξύ. Κάτι τέτοιο θα ήταν χρήσιμο, ως αυξημένη δηλαδή στρατιωτική παρουσία, γιατί η παρουσία τελικά ε, είναι ένας σπουδαστικός παράγοντας που καθορίζει το πώς κινούνται οι, οι κατατόπους σε διάφορα επίπεδα. Τώρα το Ουσμπεκιστάν, ε, λόγω της γεωγραφικής του και όχι μόνο ε, κατάστασης, θέσης, μεταφάλει και αυτό και προσαρμόζει τη δική του πολιτική σε ό,τι αφορά δηλαδή, την πολιτική του για την Κεντρική Ασία. Άρα λοιπόν, λαμβάνοντα υπόψη όλου αυτού του επιμέρου παράγοντε, και τις συνισταμένες, ε, επανέρχομαι στο κύριο μήνυμα το οποίο εγώ θεωρώ ως πολύ σημαντικό να σας ε, μεταβάσω. Είναι το ότι η πολιτική της Δύσης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την πλευρά του ΝΑΤΟ, θα πρέπει ή μέχρι στιγμής είναι, ε, έχει ε, έναν, ε, ακολουθεί μια κατεύθυνση απάντησης ή ανταπόκρισης σε όσα συμβαίνουν. Δεν έχει δηλαδή σχεδιάζει προς τα μπροστά. Το τι θα πρέπει να γίνει δηλαδή στο μέλλον δεν έχει προοπτικό χαρακτήρα. Θα πρέπει ε, δηλαδή να αξιολογηθεί καλύτερα το πώς και με ποιον τρόπο θα διαμορφωθεί η παρέμβαση της ε, Δύση ε, στο μέλλον σε όλη αυτή την περιοχή, στην Κεντρική Ασία και στο Νότιο Κάφκασο και στην μέσα, Ανατολή και ούτω καθεξής. Γιατί αυτή η διαδικασία λοιπόν σύνθεσης και αποσύνθεσης αν θέλετε δηλαδή συνένωση και κατατερματισμού συνεχίζεται και υπάρχουν διαφορετικοί διαφορετικά κέντρα, διαφορετικοί παίκτες αν θέλετε σε αυτή την ε, ε, σε αυτό, το μοσαϊκό με, διαφορετικές, με διαφορετική ατζέντα ο καθένας από αυτούς. Σε ό,τι αφορά τώρα το, ε, την οικονομική διάσταση του Αφγανιστάν, θα πρέπει ακριβώς να ενταχθεί σε αυτήν την, στον εμπορικό, στο εμπορικό τμήμα της στρατηγικής υποδομής φωτιαστικής και ούτω καθεξής. Ε, γιατί βέβαια υπάρχει και όλη αυτή η περιγνωμοσύνη που έχει συγκεντρωθεί από τους αρμοδίους για την εφοδιαστική στο στρατιωτικό επίπεδο και σε σχέση και με άλλες χώρες όπως ε, το ε, Ουσμπεκιστάν και το Τυριστάν και άλλους. Γιατί ακόμα και το Ουσμπεκιστάν είχε δηλώσει ότι παραμένει ουδέτερο, αλλά τελικά επέτρεπε τη μεταφορά μέσω της επικράτειάς του κάποιου ε, στρατιωτικού υλικού, για παράδειγμα καυσίμων. Άρα λοιπόν η διαδικασία αυτή θα στεφτεί με επιτυχία μόνο εφόσον υπάρξει ισχυρή πολιτική βούληση. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι που μόλις ανέφερα, δηλαδή το οικονομικά, αλλά και σε ό,τι αφορά γενικότερα το μέλλον του Αφγανιστάν. Και μετά το ερώτημα που τέθηκε σε ό,τι αφορά το ποιο είναι ο στρατηγικός στόχος της παρουσίας των στρατευμάτων ε, και τη διάρκεια Εντάξει, σίγουρα όταν ακούγεται ότι ε, το χρονοδιάγραμμά μας ε, τελειώνει, σε λίγο θα αποχωρήσουν τα στρατεύματα, όλα αυτά δημιουργούν περισσότερη αβεβαιότητα εκεί. Θα σταματήσω εδώ. Φαντάζομαι πως θα τεθούν περισσότερα ερωτήματα και βέβαια θα χαρώ πολύ να τα απαντήσω. Αλλά ενδεχομένω και άλλα ερωτήματα τα οποία να σχετίζονται με την ευρύτερη κατάσταση στην περιοχή. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντοροτέ Βαντάμα έχει τώρα το λόγο από, την, από το Καθολικό Πανεπιστήμιο του, της Λουβέ. Thank you very much. I would like to join my uh, fellow in, thank Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας και είναι τιμή μου να βρισκόμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Εγώ θα κάνω ένα βήμα πίσω, δηλαδή θα εξετάσω μόνο το Αφγανιστάν και θα εξετάσω λίγο την ε, ευρύτερη κατάσταση στην περιοχή. Ε, χρησιμοποιώ δηλαδή πολλού ε, χάρτε στη δική μου παρουσίαση. Ποια είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Αφγανιστάν. Η γεωπολιτική δυναμική έχει να κάνει όλο ένα και περισσότερο, υπεριστρέφεται όλο ένα και περισσότερο γύρω από το Πεκίνο και την Κίνα. Ε, και η, ε, ε, από το, γύρω από το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή ηγεσία δεν αναγνωρίζει το ρόλο των ΗΠΑ. Άρα λοιπόν υπάρχει εδώ αυξημένος ρόλος της Κίνας και της Ινδίας αλλά και οι ΗΠΑ παραμένουν εμπλεγμένες εδώ γιατί δεν θέλει να χάσει σε επιρροή. Όλα αυτά λοιπόν επηρεάζουν την κατάσταση που ισχύει αυτή την κατάσταση στο Αφγανιστάν. Πιο συγκεκριμένα ε, το Αφγανιστάν αποτελεί εδώ ένα πολύ σημαντικό σημείο, έναν άξονα λόγω ακριβώς της ευραλικής του γεωγραφικής θέσης. Και τα ευάλωτα σημεία του Αφγανιστάν έχουν ιδιαίτερε επιπτώσει όχι μόνο για την ίδια τη χώρα, αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Σα δείχνω εδώ στη διαφάνεια δύο ε, χάρτε. Βλέπετε λοιπόν πω είναι μια χώρα ενδιάμεση, αν θέλετε, σε μεγάλε δυνάμει. Ένα buffer state όπω ε, λεγότανε και στο 19ο αιώνα αργότερα, αλλά και τη σήμερα ημέρα. Και αυτό επηρεάζει την ευρύτερη ε, κατάσταση ασφαλεία. Δηλαδή, ό,τι συμβαίνει στο Αφγανιστάν αυτομάτω έχει επιπτώσει στην ευρύτερη περιοχή, ακριβώ επειδή είναι χώρα buffer. Και βέβαια πάντοτε σε αυτή την περιοχή έχουμε να κάνουμε με, δύο, με, με τρεις δυνάμεις, δηλαδή την Ινδία, το Πακιστάν, την Κίνα και τη Ρωσία που δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα. Συχνά η αστάθεια στο Αφγανιστάν χρησιμοποιείται ως μοχλός από άλλες δυνάμεις και ιδιαίτερα από το Πακιστάν γιατί αυτές οι διαπραγματεύσεις πολύ συχνά σημαίνουν ότι μάλλον η συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις αποτρέπει από το να εστιαστεί κανεί στο πυρηνικό πρόγραμμα του ιδίου του Πακιστάν. Το Πακιστάν έχει μια προσέγγιση επί των πυρηνικών που δεν συμμερίζεται τις ευρωπαϊκές ή δυτικές αρχές. Θεωρεί το Πακιστάν ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα σε οποιαδήποτε στιγμή απειλείται. Θα αναφερθώ πάρα πολύ σύντομα στι ΗΠΑ γιατί γνωρίζετε ήδη ποιοι είναι οι στόχοι των πολιτείων στο Αφγανιστάν, αλλά δεν μπορεί κανείς να δει την κατάσταση στο Αφγανιστάν χωρίς να καταλάβει και τι στοχεύσει των τεσσάρων περιφερειακών δυνάμεων που ενέχονται. Ποια είναι τα συμφέροντά του στο Αφγανιστάν και ποιο είναι ο ανταγωνισμό μεταξύ του. Πολύ σύντομα λοιπόν. Οι Ηνωμένε Πολιτείε θέλουν να αποφύγουν ένα αποτυχημένο κράτος. Που αυτή τη στιγμή είναι περίπου η κατάσταση, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι υποσυζήτηση. Οι Αμερικανοί επίσης δεν θέλουν να αφήσουν πολιτικό κενό, γιατί έχουμε δει τι σημαίνει αυτό. Δεν θέλουν και άλλη επίθεση τύπου 11 Σεπτεμβρίου αλλά δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν και το απίθαρχο, θα λέει κανείς, Πακιστάν. Η διαφάνεια αυτή νομίζω ότι δείχνει αρκετά καλά την κατάσταση της ισορροπίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Πακιστάν και το πόσο έχει ε, ε, τι αντίκτυπο έχει η κατάσταση του Αφγανιστάν επί της σχέσης. Οι Αμερικανοί αισθάνονται προδομένοι από τη στάση του Πακιστάν και το αντίστροφο. Επανερχόμενοι στο Πακιστάν, το Πακιστάν θεωρεί ότι ό,τι και να συμβαίνει στον κόσμο που να αφορά στο Πακιστάν έχει σχέση και με την Ινδία. Περνάει λοιπόν από το πρίσμα, από την οπτική και της Ινδίας και αυτό εξηγεί μεγάλο μέρος και της ε, στρατηγική του τοποθέτησης γιατί τοποθετείται έναντι τη Ινδία το Πακιστάν. Και αυτό εξαρτάται από το στρατιωτικό οικοδόμημα και όχι την πολιτική ελίτ. Η πολιτική ηγεσία μπορεί να αναλάβει ορισμένες κινήσεις εφόσον όμως δεν αποκλίνει ιδιαίτερα από το στρατιωτικό δόγμα. Οι Αμερικανοί γνωρίζουν ότι μπορεί να μιλήσει κανείς με την Ισλαμαμπάντ, αλλά τελικώς οι αποφάσει θα λαμβάνονται στο Ραγουαλπίντι, δηλαδή στην έδρα της στρατιωτική ηγεσία. Άλλο σημαντικό στοιχείο είναι τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών, τα οποία είναι ορθάνυχτα αυτή τη στιγμή, σουρωτήρι, πάει και έρχεται όποιος θέλει, αν και βεβαίω υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία από τα οποία υποτίθεται ότι πρέπει να επιτρέπεται να περνούν οι παστού μεταξύ των δύο, που κατοικούν και στι δύο δηλαδή χώρες. Οι Πακιστανοί όμως φοβούνται ότι οι Παστούν θα μπορούσαν να επιδιώκουν μια πολιτική ανεξαρτησία, μια δημιουργία ενός Παστούνιστάν. Και δεν βοηθάει και η αναγνώριση της γραμμής Ντιουράν που είναι τα σύνορα τα επίσημα μεταξύ των δύο χωρών. Το Πακιστάν επιδιώκει μια κυβέρνηση φιλική προς το Πακιστάν ή ουδέτερη. Το μέτωπο με την Ινδία είναι ανοιχτό. Όλοι γνωρίζουμε για το Κασμίρ που είναι το πιο καυτό ζήτημα μεταξύ των δύο αυτών χωρών Και αυτό σημαίνει για το Πακιστάν μια εμπόλεμη κατάσταση και με τις δύο σύνορες όμορες χώρες. Το Πακιστάν επίσης προσπαθεί να αποδυναμώσει την Ινδία από το να εγκατασταθεί στα σκύπτρα της μεγάλης πυριακής δύναμης. Δεν θέλει το Πακιστάν η Ινδία να ανακατεύεται πολύ με τα θέματα του Αφγανιστάν. Και αυτό το λαμβάνουν υπόψη οι πολιτικής, γιατί όσο η Ινδία ανακατεύεται, τόσο χειρότερη, πιο αρνητική είναι η αντίδραση του Πακιστάν. Και όταν λέω αρνητική, εννοώ υπό τη στρατηγική έννοια, με ένοπλες ομάδες που θεωρούνται καλοί αντάρτες, κακοί αντάρτες, καλοί τρομοκράτες, κακοί τρομοκράτες και και ούτω καθεξής. Τώρα εγώ συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό της διαδικασίας ε, της, της Καμπούλ, της Καμπούλ Process δηλαδή, που αναφέρθηκαν και τα άλλα μέλη του πάνελ, αλλά πρέπει να δει κανείς πώς θα αντιδράσει το Πακιστάν. Γιατί όσο οι Ταλιμπάν θα μπορούσαν να δεσδίσουν την πολιτικό σκηνικό και να έχουν δηλαδή λόγο και για την πολιτική κατάσταση στο Πακιστάν, τόσο λιγότερο λιγότερη επιρροή θα έχει το Πακιστάν επ' αυτόν. Και ίσως για αυτό το λόγο το Πακιστάν να μην είναι τόσο ανοιχτό σε αυτή την ερηφτική διαδικασία και να προσπαθήσει να την αποσταθεροποιήσει πολύ περισσότερο. Πάω τώρα στην Ινδία, η οποία είναι μια ανερχόμενη δύναμη, θέλει να συμπεριφέρεται ως τέτοια, ως μεγάλη δύναμη. Και το Αφγανιστάν είναι με καλή δίωδος για τη φιλοδοξία της, βλέπει την περιοχή ως φυσικό της δικαίωμα και θέλει και να αντισταθμίσει την επιρροή της Κίνας. Διότι ως γνωστόν επίσης, η Κίνα και η Ινδία αντιπαλεύουν για την ε, συνολική ηγετική θέση της περιοχής. και υπάρχει και η απειλή ε, τρομοκρατικών επιθέσεων από το έδαφος ε, του Αφγανιστάν στο έδαφος Ινδίας. Μια περαιτέρω σταθεροποίηση ασφαλείας και οικονομική θα μπορούσε να εξεταστεί για την Ινδία η οποία έχει κάθε συμφέρον στο να σταθεροποιήσει την κατάσταση, να βοηθήσει σε μια σχετική ειρήνευση. Η δε Κίνα έχει τρεις στόχους. Θέλει να ενισχύσει την κεντρική της ισχύ, δύναμη, εξουσία, ε, με κόκκινο στο χάρτη βλέπουμε την περιφέρεια την πιο κοντινή, την Σιντσέγκ. η οποιαδήποτε έλλειψη σταθερότητα στο Αφγανιστάν έχει αντίκτυπο στην περιφέρεια αυτή την κινέζικη, η οποία έχει σημαντικό μουσουλμανικό στοιχείο στον πληθυσμό της. Επομένως η Κίνα έχει επίσης συμφέρον σταθεροποίησης, ώστε να μην έχει διείσδυση από Ισλαμικές τρομοκρατικές ομάδες στο έδαφος της. Και κάτι ακόμα που είναι σημαντικό για την Κίνα είναι η ανάπτυξη του νέου δρόμου του μεταξιού η οικονομική ανάπτυξη χάρη εσωτερική σταθερότητα δηλαδή για την Κίνα και η όποια έλλειψη σταθερότητα στο Αφγανιστάν δεν θα τη βοηθήσει να ολοκληρώσει την υποδομή ή το στόχο αυτό. Και για το λόγο αυτό είναι υπέρ της σταθεροποίησης. Επίσης, βέβαια, προσπαθεί και η Κίνα να αντισταθμίσει την επιρροή της Ινδίας. Πολλοί αναφέρθηκαν σε επένδυση σε στρατιωτική βάση στο Αφγανιστάν ο πλευράς και επομένως θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι και η στάση της Ινδίας και αντίστροφα. Και θα ήθελα να κλείσω με αυτά που θεωρώ ότι πρέπει να είναι τα σημεία που πρέπει να προσέξει κανείς για το μέλλον του Αφγανιστάν. Πρώτα απ' όλα, ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι πώς η Ινδία θα αυξήσει ή όχι την επιρροή της, το ρόλο της στο Αφγανιστάν. Πώς αυτό θα έχει αντίκτυπο επί της εξωτερικής πολιτικής της, του Πακιστάν και πώς αυτό θα επιδράσει στους Ταλιμπάν θα τους απομακρύνει από την ειρηνευτική διαδικασία. Θα υπάρχουν και άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις κατά της Ινδίας, ώστε η Ινδία να εστιάζεται σε αυτές και όχι στο Αφγανιστάν. Βεβαίως και η κατάσταση στο Κασμίρ έχει δυνητικά αποσταθεροποιητικό ρόλο και επιρροή. γιατί θα μπορούσε να επηρεάσει απευθείας το Αφγανιστάν και υπάρχουν και οι αντιπαραθέσεις διαντιπροσώπων που διεξάγονται μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν ή μάλλον Ινδίας και Κίνας γιατί δεν αντιπαρατίθενται ευθέω, αλλά σε άλλα μέτωπα υπάρχει η κατάσταση με τη Βόρεια Κορέα, υπάρχει η Βόρεια Κινέζικη θάλασσα, για την Ινδία υπάρχει η Σρι Λάνκα, υπάρχει το Πακιστάν. Αλλά μία κάποια προσέγγιση των τελευταίων ετών μεταξύ επίσης Ινδίας και Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορούσε να είναι αποσταθεροποιητικός παράγοντα γιατί η Κίνα θα μπορούσε να επιθυμήσει την ε, αποσταθεροποίηση τη Ινδία μέσω του Πακιστάν. Βεβαίω η συμφωνία του 2006 για τα πυρηνικά μεταξύ Ινδία και Ηνωμένων Πολιτειών νομίζω ότι είχε χαρακτηριστεί ω προδοσία, αν δεν κάνω λάθο, από τους Πακιστανούς οι οποίοι θεώρησαν ότι αυτό ήταν πισόπλατο μαχαίρωμα από πλευρά των Αμερικανών. Άρα πρέπει να δει κανείς και πώς αυτή η προσέγγιση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ινδίας επιδρά. Αλλά και η Ινδία έχει κάθε συμφέρον να επενδύσει στη σταθερότητα και την ειρήνευση της περιοχής. Άλλο θέμα που πρέπει να δει κανείς είναι τα εσωτερικά ύδατα, τις πλωτές οδούς, το εμπόριο, τις επενδύσεις που θα μπορούσαν να είναι παράγοντες καλύτερης συνεργασίας και σταθεροποίησης. Επίσης οι μεταναστεύσεις, οι μεταναστευτικές ροές. Οι εμπορικές επενδύσεις και οι μεταναστευτικές ροές θα μπορούσαν να είναι θύρες, δίωδοι, για μία κάποια γεφύρωση των διαφορών Ινδίας και Πακιστάν, έχοντας και εταίρους που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τα θέματα μετανάστευσης. Αλλά θα ήθελα να κλείσω θετικά λέγοντας ότι ο ανοιχτός πόλεμος μάλλον θα αποφευθεί. Η Κίνα και η Ινδία δεν θα πάνε σε πόλεμο. Δεν νομίζω ότι θα πάνε σε πόλεμο, λέει ο Μιλήτρια. και η Ουάσιγκτον παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την οποιαδήποτε πυρηνική κλιμάκωση. Οι Αμερικανοί θα αντιδρούσαν πάρα πολύ γρήγορα όπως αν στο παρελθόν σε οποιαδήποτε τέτοια κλιμάκωση. Μάλιστα λέει ο Πρόεδρος, θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στα μέλη για την γενική συζήτηση, ο κύριος Ντανζό, καταρχάς. ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. συμφωνώ με τον κύριο Τιπάλο, θα πρέπει να αποφασίσουμε, να αποφύγουμε συγγνώμη, τον κινησμό για το Αφγανιστάν, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει κάποιος σκεπτικισμό σε σχέση με αυτά που άκουσα όσον αφορά τις δικές μας τις συμβολές. Να επανέλθω σε κάποια απλά πράγματα. Γιατί πήγαμε στο Αφγανιστάν. Πήγαμε εκεί γιατί είχαμε την Αλκάιντα και όχι τους Ταλιμπάν δεν κάνουν την παρέμβαση λόγω των Ταλιμπάν, αλλά λόγω της Αλκάιντα. Μετά τη στρατιωτική νίκη λοιπόν θεωρήσαμε ότι θα επιβάλαμε την δημοκρατία όπως την Σουηδία και την Ελβετία και στο Αφγανιστάν. Αλλά αυτό δεν συνέβη και σήμερα είμαστε παγιδευμένοι σε μια τέλειωτη σύγκρουση και προσπαθούμε να βρούμε ένα διέξοδο. Κάτι το οποίο όμως δεν με πείθει εδώ ως λύση. Είμαστε βέβαιοι ότι αν δεν υπάρχει η Αλκάντα, οπωσδήποτε υπάρχει το Ισλαμικό κράτος στο Αφγανιστάν. Μάλιστα είχαμε και μια τρομακρατική ενέργεια με 20 νεκρούς στην Καμπούλ που ανέλαβε την ευθύνη το Ισλαμικό κράτος αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση πια. Έχουμε λοιπόν περισσότερε τρομοκρατικέ ομάδε από ό,τι όταν κάναμε την παρέμβαση και έχουμε του Ταλιμπάν που ελέγχουν περισσότερο έδαφο σε σχέση με την κορύφωση της δικής μας στρατηγικής παρουσίας. Και εδώ ακούω ότι του χρόνου θα πάνε τα πράγματα καλύτερα επειδή οι Ταλιμπάν θα καταλάβουν ότι υπάρχει, ότι δεν θα υπάρχει διέξοδο στρατιωτική. Αλλά συγγνώμη, αυτό τον καταλάβει εδώ και καιρό είναι ανόητη. Πώ θα καταλάβουν λοιπόν οι Ταλιμπάν του χρόνου ότι δεν υπάρχει διέξοδο στρατιωτική αν δεν το έχουν ήδη ε, καταλάβει με την παρουσία 150.000 ανδρών δυτική στρατιωτικής δυναμής. Αν με τόσου άντρε δεν, δεν το είχαν καταλάβει, τι να πω. Το πρόβλημα είναι πολιτικό. Το θέμα είναι να καταλάβουμε τι επιθυμούν, τι θέλουν οι Ταλιμπάν. Θέλουν να καταλάβουν την εξουσία, θέλουν να τη μοιραστούν δεν ξέρω. Θα ήθελα να ακούσω εδώ κάποιες απαντήσεις, έτσι, γιατί αυτό το σημείο κλειδί, γιατί το να κάνουμε εικασίες ότι θα, ότι θα, προ, θα προκαταβάλουν το ενδεχόμενο στα ειδική κτλ. Δεν ξέρω αυτή η επίγνωση για ποιο λόγο θα πρέπει να γίνει του χρόνου και όχι μέχρι τώρα με 105.000 ε, άντρες στατιωτική δύναμη από τη Δύση. Θέλω λοιπόν να υπάρχει περισσότερη εδώ λογική σε σχέση με το τι αναμένουμε από τις κινήσεις των διαφόρων πολιτικών παραγόντων. Για να καταλάβουμε κατά πώς θα υπάρξει μια διέξοδος ε, αποτελεσματική ή γρήγορη σε αυτή την σύγκρουση και αυτή τη μεγάλη πολιτική, την υψηλή πολιτική, εγώ δεν την καταλαβαίνω. Δηλαδή ο τόπος όπου όλα τα συμφέροντα τα δυτικά συγκλίνουν, αυτό το καταλαβαίνω είναι στρατηγική η γεωγραφική θέση του Αφγανιστάν εντάξει σε σχέση με τις γειτονικές χώρες όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι μου φαίνεται ότι κάποιες μεγάλες δυτικέ χώρες ασχολούνται με τις σχέσεις τους με την Κίνα, τη Ρωσία και άλλες χώρες άσχετα με το τι συμβαίνει με το Αφγανιστάν. Ίσως να είναι καλό αυτό ή κακό, δεν ξέρω. Ίσως να το πληρώσουν αυτό ή όχι, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι δεν θα πρέπει να κρίνουμε τη σχέση μας με αυτό το τμήμα του, κόσμου, σύμφωνα με αυτό που συμβαίνει στο Αφγανιστάν. Δεν είναι ευχάριστο, αλλά δεν νομίζω είναι και τόσο σημαντικό αυτό το θέμα του Αφγανιστάν. Έχουν επενδυθεί μεγάλα κεφάλαια σε σχέση με το Αφγανιστάν μας ενοχλεί ίσως, αλλά πολλές χώρες νομίζω ότι πια επιθυμούν να αποσυρθούν, να φύγουν από εκεί. Γιατί έχουμε τάση να λέμε ειδήσει και κλπ. Όχι, δεν ισχύει. Αν έρθετε στο Παρίσι, που δεν είναι μικρή πρωτεύουσα μικρή χώρα, έτσι, όσον αφορά στρατιωτικέ ε, επιχειρήσει, θα σα πει ο ηγέτη ότι Εντάξει, είναι μεγάλη προτεραιότητα για μα το Αφγανιστάν, αλλά ίσω αυτό να είναι λάθο. γιατί εδώ και 17 χρόνια η κατάσταση δεν εξελίσσεται. Θα πρέπει λοιπόν, αν χρειαστεί να στείλουμε στρατιωτικέ δυνάμει, θα πρέπει να εξηγήσουμε στου πολίτε γιατί στέλνουμε στρατιώτε, γιατί πάμε να πολεμήσουμε εκεί, γιατί δεν του αρέσει. Αν στέλνουμε λοιπόν εκεί στρατιώτε. Ελπίζοντα ότι πολεμώντα του Ταλιμπάν θα έχουμε ιστορική δύναμη, αυτό νομίζω ότι είναι ψευδέστηση. Συγγνώμη, δεν θέλω να σας χαλάσω τις ψευδεστήσει, αλλά έχω πολλές αμφιβολίε. Και δεν βλέπω κάτι που να μου τις διασκεδάζει. Και το θέμα με το Πακιστάν και την Ινδία είναι πολύ πιο σοβαρό σε σχέση με και δεν είμαι τόσο βέβαιο όσο εσεί ότι μπορεί να συμβεί κάτι πολύ σοβαρό μεταξύ Πακιστάν και Ινδία. Έχουν παρουσία οι Πακοί στο Πακιστάν, λέτε, και θα ασχοληθούν. Πώ, πώς. Εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτό δεν ισχύει. Και δεν τους νοιάζει και τόσο τους ε, Πακιστάνους ηγέτες το τι μπορούν να κάνουν οι Αμερικανοί. Πάντως, να θεωρήσουμε ότι μια σύγκρουση μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας θα μπορούσε εύκολα να επεκταθεί, επειδή πολύ μεγάλες δυνάμεις ενδιαφέρονται, τότε, τι να σας πω, εμένα δεν με πείθει αυτό. Θα ήθελα να συμφωνήσω, αλλά δεν βλέπω τίποτα στα γεγονότα του Αφγανιστάν να μας οδηγούν σε αισιοδοξία. Thank Ευχαριστώ, κυρία Λουζίν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν συμβαίνει συχνά, αλλά αυτή τη φορά μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα με τα όσα μόλις είπε ο κύριος Ντόμσον. Δεν θέλω δηλαδή τώρα να τονίσω ιδιαίτερα κάποια προοπτική, αλλά πραγματικά ε, που άκουσα αυτές τις παρουσιάσεις ε, θυμήθηκα μια αυτοβιογραφία μιας νεαρής ε, Αφγανής με τον τίτλο «Μόνο για κλάματα ανακατάσταση». ε, Δηλαδή, λαμβάνοντα υπόψη όλε τι διαφορετικέ στρατιωτικέ εναλλακτικέ, ε, δεν διαπιστώνω κανεί να ασχολείται ή ασχολούνται όλοι όλο ένα και περισσότερο με το τι συμβαίνει ακριβώς στους ανθρώπους αυτής της χώρας, ε, ποια είναι η ζωή τους, ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσης. Τώρα, θα ήθελα να θέσω κάποια πιο συγκεκριμένα ερωτήματα. Αναφέρθηκε επανειλημμένα το ζήτημα της μετανάστευσης. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα ειδικότερα προς την υπηρεσία εξωτερικής δράσης τι ακριβώς εννοεί όταν λέει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας ε, ε, συνεργασίας θα υπάρξει αυξημένη συνεργασία σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση. Δηλαδή τι, περισσότερες απελάσεις Αφγανών προς το Αφγανιστάν, για παράδειγμα από τον Frontex, από, δηλαδή ε, άτομα τα οποία βρίσκονται στην Γερμανία ή στην Αυστρία ή στη Σουηδία. Ε, μόλις τώρα μας περιγράψατε λεπτομερώς την κατάσταση ασφαλείας στο Αφγανιστάν. Ε, και βέβαια λαμβάνοντα υπόψη αυτή την κατάσταση, πώ μπορούμε να προβούμε σε μια τέτοια πελασία σε αυτή τη χώρα πρόλευση. Από εκεί και μετά, σε ό,τι αφορά την, ε, ε, το, το κατά πόσο τίθεται προποθέσει για την χορήγηση ανθρωπιστική βοήθεια, σε ό,τι αφορά ακριβώ αυτέ τι τις επιστροφές, αυτές τις Τώρα, ο ρόλος αυτής της συνεργασίας ε, με τον ε, Ταλιμπάν δεν ξέρω πώς αξιολογείται, ασχέτως του δηλαδή τελικά αν θα ε, εφαρμοστεί ή θα πετύχει στην πράξη όχι. Κάτι τέτοιο δηλαδή έρχεται σε αντίθεση με την στρατηγική των, των ΗΠΑ εκεί ή όχι. Ο κύριος Αστροβίτσιος μας είπε ότι στο στρατιωτικό βέβαια το κάνουμε αυτά και αυτά, ενώ στο μη στρατιωτικό κάνουμε εκείνα. δεν μπορώ να φανταστώ ότι έχουμε να κάνουμε εδώ δηλαδή με δύο τμήματα στρατηγικής τα οποία αντίκειται στο ένα στο άλλο, είναι αντιφατικά. Ενώ ο κύριος Αντιστροβίτσιος είπε επίσης ότι δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για τους Ταλιμπάν γιατί είναι μια σειρά από διαφορετικές ομάδες εδώ οι οποίες δραστηριοποιούνται. Ενώ από την άλλη αναφέρεται ότι υπάρχει συνεργασία με τους Ταλιμπάν. Τελικά μπορούμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας μια τέτοια προσέγγιση. Και αυτή η προσέγγιση πραγματικά τελικά μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής, ναι ή όχι. Γιατί νομίζω πως μερικές ε, φορές ε, έχω την εντύπωση ότι αυτό που συμβαίνει είναι απλώς ε, ένα brainstorming. Ο καθένας έχει τη δικιά του ιδέα και λέει ας κάνουμε αυτό, ας κάνουμε εκείνο, χωρίς να υπάρχει συντονισμός. Ε, παλαιότερα εδώ είχαμε και εκπροσώπους από την πλευρά της Αφγανικής κυβέρνησης όταν κάναμε συζητήσεις σε σχέση με το Αφγανιστάν. Αυτή η, θέση τώρα του Πρόεδρου σε ό,τι αφορά τη, την αύξηση των στρατιωτικών δυνάμεων τώρα του ΝΑΤΟ θα επηρεαστεί δηλαδή η σχέση του Πρόεδρου με την, ε, με την ε, Δύση. Έχουν γίνει συγκεκριμένα σχέδια δηλαδή και έχει υπάρξει κάποια συνεννόηση σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έλσεν από την ε, προσωπία στο Αφγανιστάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τις παρεμβάσεις τους. Θα είμαι σύντομος, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. παρακολούθησα πολύ προσεκτικά την παρέμβαση του συναδέλφου των Ζων αλλά και τη ε, Γερμανίδα συναδέλφου. Ζητώ συγγνώμη, δεν έχω τα γυαλιά μου, οπότε δεν καταφέρατε να διαβάσω το όνομά τη. Συμφωνώ λοιπόν και συντάσσω με τα ερωτήματα ε, του συναδέλφου των Ζων αλλά και τη Γερμανίδα συναδέλφου. Και να πω ότι εγώ ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη στρατηγική εξόδου από το Αφγανιστάν, το exit strategy. Εάν υπάρχει μια τέτοια στρατηγική, πώς διαμορφώνεται και πότε μπορούμε να αναμένουμε τα πρώτα βήματα στο πλαίσιο αυτή τη στρατηγική για την έξοδο του Αφγανιστάν. Uh, ευχαριστώ. Επειδή δεν επιθυμεί κάποιο άλλο το λόγο, να κάνω κι εγώ κάποιε ερωτήσει. Και αυτή την προσφορά και το πρόεδρο κάνει Νομίζω ότι όλοι ήμασταν θετικοί για αυτό το θέμα. Οπότε σας παρακαλώ να επικεντρωθείτε τώρα σε θέματα όπως η εκλογική διαδικασία γιατί εδώ δεν χωρούν συναισθηματισμοί, πρέπει να συζητήσουμε θέματα σταθερότητας. Βεβαίω υπάρχουν προφανείς προκλήσεις σε αυτή τη δικασία. Μπορείτε να μας το αναπτύξετε περισσότερο αυτό. Δηλαδή, τι απόψε έχετε αυτή την συγκεκριμένη διαδικασία. Διακόπτη πρόεδρος. Ναι, παρακαλώ. Ναι, μία μικρή ε, προσθήκη θα ήθελα να κάνω στο προηγούμενο ερώτημά μου, γιατί το θυμήθηκα τώρα. Αναφέρθηκε πως η κατάσταση σε ό,τι αφορά το ΝΑΕΣ, ε, το Ισλαμικό κράτος δηλαδή και του Ταλιμπάν είναι πολύ περίπλοκη. Δηλαδή, ποια ακριβώς είναι η σχέση μεταξύ τους, ISIS και Ταλιμπάν. Μπορούμε να λάβουμε περισσότερες εξηγήσει με την ίδια σειρά ο κ. Κλίσσερ πρώτα. Ευχαριστώ για αυτές τις ερωτήσεις. Πρώτα, η ερώτηση της κ. Λέζινγκ για τη μετανάστευση. Που είναι πολύ σημαντικό θέμα. Υψηλά στο θεματολόγιο των επαφών με τους οργανούς και όπως είπατε, είναι τμήμα της συμφωνίας εταιρική σχέση και συνεργασία που υπογράψαμε πέρσι μεταξύ της είπα της εκπροσώπου και της αυγανικής κυβέρνησης. Ο διάλογος για τη μετανάστευση δομείται και διοργανώνεται μέσω του CEPD, αλλά η συνεργασία με το Αυγανιστάν εν μέσω του Joint Way Forward είναι, συγγνώμη, μία μη νομικά δεσμευτική συμφωνία που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Αφγανιστάν για την παράνομη μετανάστευση. Δηλαδή, είναι η συνεργασία που δεν αφορά τους μετανάστες, αλλά αφορά αυτούς που προσπαθούν να εισέλθουν στην ΕΕ παράνομα και έχουν εξαντλήσει όλα τα νομικά τους μέσα για παραμονή στην Ένωση και έχουν απορριφθεί. Συμφώνησε λοιπόν το Αφγανιστάν να αποδεχτεί αυτές τις πτήσεις επιστροφής επαναπατρισμού αυτών των ατόμων που διοργανώνουν οι χώρες μέλη και η Frontex. Αφορά λοιπόν αυτού που δεν διαθέτουν το νομικό Καθεστώ για παραμονή στην Ευρώπη και γνωρίζουμε τις συζητήσει που σχετίζονται με τα θέματα ασφάλεια. Τώρα, ο επαναπατρισμός αυτών των ατόμων στο Αφγανιστάν ή στην Καμπούλ είναι ένα θέμα όπου προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τις χώρες μέλη να κάνουμε μια καλύτερη αξιολόγηση της κατάστασης η οποία μεταβάλλεται συνεχώς παντού στο Αφγανιστάν. Από μόνη της δεν είναι απειλητική για τη ζωή αυτή η κατάσταση σε όλο το Αφγανιστάν. Όμως θα πρέπει να δούμε προσεκτικά τις διάφορες καταστάσεις και θα πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες μέλη ώστε στα πλαίσια των δικών τους διαδικασιών ασύλου να κάνουν τις απορρίψεις εκεί που χρειάζεται. Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ παροχής ανάπτυξης βοήθειας στο Αυγανιστάν και το Αυγανιστάν να αποδεχτεί τον, τους επαναπατρασμούς αυτούς. Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο θεμάτων. Ίσως θα πρέπει να πω και δύο λόγια σε σχέση με το επιπλέον ερώτημά σας για, την, για τον ΤΑΕΣ και τους Ταλιμπάν. Είναι κάπως περίπλοκη αυτή η σχέση και είναι αλήθεια ότι υπάρχουν τοπικές ομάδες και Ταλιμπάν και ΤΑΕΣ που πολεμούν συμπολεμούν και συνεργάζονται σε κάποιες περιοχές, σε άλλες όμως είναι αντιμαχόμενες. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να διακρίνει κανείς τα συμφέροντα. Και εξαρτάται πάρα πολύ αυτό από τη τοπική δυναμική εξουσία και τις τοπικές διαμάχες. Κάποιες ομάδες ένοπλες ε, το θεωρούν ως ευκαιρία για να κερδίσουν έδαφος σε θέματα τακτικής. Δηλαδή συμμαχούν για να πολεμήσουν καλύτερα τον τακτικό στρατό του Αφγανιστάν. Και αυτό ακριβώ εννοώ ότι είναι περίπλοκη η σχέση. Δηλαδή είναι δύσκολο κανεί να κατανοήσει και να προβλέψει τη δυναμική ή τι δυναμικέ μεταξύ των ε, ενόπλων ομάδων στο Αφγανιστάν. Θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Ντιπάολο έχει το λόγο. Ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις σας. Και βέβαια δεν πρέπει ποτέ να συγχαίουμε τον σκεπτικισμό ή την προσοχή με τον κινησμό. Καλό θα ήταν όλοι να είμαστε πιο προσεκτικοί και αν ε, επανέλθουμε στην εποχή πρώτου 2001 θα έπρεπε να ξαναδούμε με σκεπτικισμό την απόφαση του να εισέλθουμε στο Αφγανιστάν. Ίσως να υπήρχαν και άλλοι τρόποι, αλλά τέλος πάντων αυτό συνέβη. Να πω το εξής για τα 16 χρόνια που είμαστε εκεί. Η σκληρή αλλά δίκαιη παρατήρηση ότι φαίνεται σαν να γλύφουμε το δάχτυλό μας για να δούμε πού φυσάει ο αέρας είναι περίπου δίκαιη. Ή ακούγεται δίκαιη. Παρότι είμαστε 16 χρόνια, ακολουθούμε μία συγκεκριμένη στρατηγική κατά της εξέγερσης από το 2008 μόνο, 8 με 9. Δηλαδή 8 χρόνια μόνο επιθετικά ακολουθούμε αυτή την τακτική που σημαίνει 8 αντί για 16 δεν είναι και τόσο παρηγορητικό αλλά τουλάχιστον βλέπουμε κάποιες ενδείξεις ότι τροποποιείται η στρατηγική όταν δεν λειτουργεί. Και στην ουσία μόνο από το τέλος του 2014 είμαστε πλέον σε μια κατάσταση ότι είναι όπου ε, έχουμε, αντιμετωπίζουμε μια καθαρά αυγανο-αυγανική υπόθεση, λέει ο μιλητής. Και πραγματικά πιστεύω ότι φτάνουμε σιγά σιγά πιο κοντά σε κάτι που φαίνεται να λειτουργεί. Αλλά πάντα είναι σωστό και κατάλληλο να αμφισβητεί κανείς τη στρατηγική. Το κατά πόσον η στρατιωτική τακτική έχει συντονιστεί με τη διπλωματική προσπάθεια, με το πολιτικό πλαίσιο. Εγώ εδώ να σας πω ότι δεν εκπροσωπώ τις ΗΠΑ αλλά το ΝΑΤΟ, αλλά οι Αμερικανοί μπήκαν εκεί με στρατηγικούς στόχους που δεν αποδείχθηκαν καθόλου ε, αποτελεσματικοί και με συμπληρωματικούς στόχους που επίσης χτίσαμε ένα σωρό κτίρια που είναι εγκαταλειμμένα. Αλλά ο στρατηγός Νίκολς έχει μια καθαρή στρατηγική αυτή τη στιγμή που την υποστηρίζει το ΝΑΤΟ με μια καλά συντονισμένη σειρά μέτρων, στρατηγική πίεση διπλωματική πίεση και κοινωνική πίεση όχι μόνο επί των Ταλιμπάν αλλά και επί της κυβέρνησης του Αφγανιστάν και των γειτόνων ώστε όλοι να εξωθηθούν προς κάποιο είδους συμφιλίωση. Έχουμε γίνει και πιο σοφιστικέ στην ε, ικανότητά μας να συντονίζουμε την πολιτική και κάτι πολύ σύντομο επί των εμποδίων που υπάρχουν, γιατί βέβαια δεν θέλω να αναφερθώ πάρα πολύ ανοιχτά στις προκλήσεις, αυτό που με ανησυχεί είναι η πολύ κακή επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης κάνει προς το εσωτερικό της χώρας του, για ότι κάνουμε την ειρήνη. Την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκα με εκπροσώπους του μεγαλύτερου τηλεοπτικού δικτύου και του ρώτησα τι κάνει ο Πρόεδρος για να επικοινωνήσει την πολιτική του στον κόσμο, μου τίποτα. Επίσης ανησυχώ όταν ακούω ότι η Δύση είναι τόσο απελπισμένη για την ειρήνη που θα την αποδεχθεί υπό οποιουσδήποτε όρους. Δεν ισχύει. Έχουμε δει από την εμπειρία στο Βιετνάμ και στην Κολομβία πόσο δύσκολο και επικίνδυνο είναι να εγκαθιστούμε ασφαλείς ζώνες, γιατί συνήθως οι ένοπλες ομάδες απλά τις χρησιμοποιούν για να επανεξοπλιστούν, να δυναμώσουν και να έρθουν ακόμα πιο επιθετικοί την επόμενη φορά. Και για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, ο ρυθμός δαπανών ασφαλείας και άλλων στον Αφγανιστάν δεν είναι βιώσιμος. Να κλείσω με αυτό. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ε, οι διερμηνείς μας θα πρέπει να μας αφήσουν έξι και μισή, λέει η Πρόεδρος, οπότε Πρέσβη Κουτέλια και κυρία Βαντάμ θα πρέπει να μοιραστείτε αυτά τα πέντε λεπτά που μας απομένουν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Πρώτα απ' όλα να απαντήσω σε αυτή την ε, τοποθέτηση σκεπτικισμού. Βεβαίως και είναι καλοδεχούμενος ο σκεπτικισμός όταν έχουμε πάρα πολλά κινούμενα μέρη σε ένα ευρύτερο πάζλ με μια κατάσταση έδαφος που αλλάζει διαρκώς είχε δοθεί ως αρχική αιτία της εμπλοκής του Αφγανιστάν η Αλκάιντα, μετά η Ταλιμπάν και τα λοιπά. Πράγματι, αλλάζει συνεχώς η, εικόνα. Όταν οι Αμερικανοί ενεπλάκησαν στην Ευρώπη, η αρχική πρόθεσή τους ήταν να καταπολεμήσουν τους Ναζί, μετά τους Σοβιετικούς και τα λοιπά. Δηλαδή ο κόσμος αλλάζει, διαρκώς, είναι διαφορετικός από αυτό που ήταν πριν από 16 χρόνια σήμερα ο κόσμος και από αυτό που ήταν πριν από 10 χρόνια. Και πριν από 10 χρόνια ήταν ε, δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι θα κατονομάζαμε τη Ρωσία στον υπαριθμόν ένα εχθρό του ελεύθερου κόσμου, ενώ σήμερα αυτό δηλώνουμε ως ΝΑΤΟ Έχουμε κρατικού και μη κρατικού φορείς και οντότητε που δρούν για διάφορες στα πλαίσια διαφόρων πολιτικών στοχεύσεων. Επομένως και ο ελεύθερος κόσμος, ξαναλέει ο μιλητής, θα πρέπει να συντονιστεί κατά τέτοιων ενεργειών. Η μεγαλύτερη μου ανησυχία, Πρόεδρε, είναι να έχουμε πολιτικές ασυντόνιστες, αντιφατικές, που να πηγαίνουν η καθεμία προς την κατεύθυνσή τους. Που έχει σχέση βεβαίως και με τις εσωτερικές πολιτικές ε, καταστάσεις στην κάθε χώρα και τον κύκλο εκλογών, αλλά ε, θα έπρεπε να εξηγήσουμε καλύτερα ποιο είναι το κόστος, ποιο είναι το τίμημα της μη ανάληψης δράσεως. Και έχουμε παραδείγματα και στη Συρία και στο Ιράκ και με ανθρώπινες ζωές, αλλά και οικονομικής ε, απώλειας. Σας ευχαριστώ. Κυρία Βαντάμ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, λέει η κυρία Βαντάμ. Η περιφερειακή προοπτική του Αφγανιστάν ε, λέει ότι ό,τι συμβαίνει στο Αφγανιστάν έχει περιφερειακό αντίκτυπο. Είτε πάει κάπου αυτή η ειρηνευτική διαδικασία είτε όχι, θα έχει αντίκτυπο στην, στον περιφερειακό σχετισμό δυνάμεων στην περιοχή. Συμφωνώ μαζί σας λοιπόν ότι ε, η αντιπαράθεση Ινδίας και Πακιστάν είναι πολύ πιο σημαντική από, την, ε, από τα πλαίσια της εξέτασης του Αφγανιστάν διότι είναι και οι δύο πυρηνικές δυνάμεις. Αυτός είναι ο λόγος. Τώρα Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για, για, για ποιον λόγο δεν θα έμπαιναν σε άμεση αντιπαράθεση αυτέ τι δύο χώρε, αλλά δεν πιστεύω ότι, ότι είναι έτσι τα πράγματα. Πάντως, οι Ταλιμπάν είναι εξαιρετικά διαφοροποιημένοι ως στη δράση τους. Οι πιο εξτρεμιστικές τους ομάδες δεν θα συμφωνήσουν στην ειρηνευτική διαδικασία. Ο πρόεδρος Γκάνη είπε ότι αυτή η ειρηνευτική διαδικασία μπορεί να προχωρήσει εφόσον γίνει σεβαστή στα πλαίσια του σημερινού συντάγματο, κάτι το οποίο δεν αποδέχονται πάρα πολλέ ομάδε των Ταλιμπάν. Και υπάρχουν και άλλε αρνητικέ επιδράσει. Η ΝΤΑΕΣ είναι μία από αυτέ τι ε, δηλητηριώδει επιδράσει επί τη ειρηνευτική διαδικασία. Ελπίζω να σφάλω, αλλά δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξη για την ειρηνευτική αυτή διαδικασία. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Θα ευχαριστήσω όλα τα αξιότιμα μέλη του πάνελ. Να τους χειροκροτήσουμε, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλα τα μέλη για τις δικές τους παρατηρήσεις και παρεμβάσεις και βεβαίως, λέει η Πρόεδρος, πολύ ευγενικά, τους διερμηνείς για το εξαιρετικό τους έργο. Εμείς Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, αύριο 9 η ώρα ακριβώς το πρωί ξεκινούμε.